Ξεκινάμε. Λιγότεροι μεν, καλύτεροι δε. Σημείο 13 της ημερήσης διάταξης. Κατάσταση στον κλάδο της με μελισσοκομείας. Κατά τη διάρκεια του 10 η Επιτροπή μα ενέκρινε ένα αίτημα προφορική ερώτηση, για υποβολή προφορική ερώτηση για την κατάσταση στον κλάδο τη μελισσοκομεία. Θα εξετάσουμε τώρα ένα σχέδιο ψηφίσματο που συνδέεται με αυτή την προφορική ερώτηση χάρη στι συνεισφορέ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Παρότι την, τον Ιούλιο η Επιτροπή αύξησε τον ετήσιο προπολογισμό για μέτρα υπέρ των μελισσουργών, παραμένει γενικευμένη ανησυχία σε ό,τι αφορά τι πολλέ προκλήσει και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδο και που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το εγγύ μέλλον, μεταξύ των οποίων οι συνθήκε παραγωγή και προώθηση. Η μεγάλη παράταση, η μεγάλη μείωση των τιμών και οι δυσκολίες λόγω της αυξανόμενης θνησιμότητας των μελισσών. Γι' αυτό το λόγο η πρόταση ψηφίσματος που υποβάλλουμε, που θέλουμε να υποβάλουμε στην Κομισιόν, ζητά να υπάρξει δέσμευση για τη διαφύλαξη και προάσπιση αυτού του πολύ σημαντικού κλάδου της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Κλάδου, ένας κλάδος όπως αυτός είναι στρατηγικός και σε ό,τι αφορά τις οικονομικές του επιπτώσεις όσο και την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την διατήρηση της βιοπικιλότητας. Άλλωστε, το έτος βιοπικιλότητας είμαστε. Μεταξύ των βασικών ερωτημάτων προς την Επιτροπή που περιλαμβάνονται στην πρόταση ψηφίσματος σας αναφέρω εντάχει να υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση μετά την λήξη των εθνικών προγραμμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αυτές προκλήσεις και τα προβλήματα του τομέα, δεσμεύσεις ε, για μια βελτίωση των στατιστικών δεδομένων και στοιχείων ε, για τον κλάδο, ιδίως ό,τι αφορά τις εξοκοινωτικές ε, εισαγωγέ μελιού που φτάνουν στην Ευρώπη δηλαδή, τη συμπερίληψη των ε, ασθενειών των ε, μελισσών μεταξύ των ε, ασθενειών που πρέπει να καταπολεμηθούν, την αντιμετώπιση της μίζωνος, της αύξησης της θνησιμότητας των μελισσών, μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη στον τομέα της κατάρτισης και ιδίως έναν νέο ρόλο ε, της Επιτροπής των κλάδο μετά το 2011. Αυτά είναι τα σημεία που υποβάλλουμε μετά από τις ε, θέσεις των διαφορών ομάδων. Πρώτα πρώτα θα δώσω το λόγο στην κυρία Λούλινγκ που είχε ζητήσει πρώτη να ξεκινήσουν αυτές οι προφορικές συζητήσεις. Ακόμα νωρίτερα ωστόσο θα ήθελα να ακούσουμε την άποψη της Επιτροπής διότι η Επιτροπή έχει κάποιες ε, καινοτομίες, κάποια γενναία στοιχεία. Οπότε θα ξεκινήσουμε μετά τη συζήτηση, αφού ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Κύριος Λαντομάντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι κάνει η Επιτροπή στον κλάδο, ιδίω την υγεία των μελισσών. Καταρχάς, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η Επιτροπή σύστησε μια διπηρεσιακή ομάδα μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων που εμπλέκονται στο θέμα. Ένα, μια ομάδα που συντονίζει η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών που θέλει να εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό. Και αυτό είναι σε ευθεία γραμμή με πρόσφατο ψήφισμα του Κοινοβουλίου που ζητά ακριβώ να βελτιωθούν οι σχέσει ε, μεταξύ των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη, τις που σχετίζονται με τις ε, ε, Το πρόβλημα της θρησιμότητας των ε, σμηνών, κάτι που έχει ήδη ζητηθεί και συζητηθεί περίπου δύο χρόνια πριν. Είχαμε ξεκινήσει μια μελέτη τότε και είχαμε ζητήσει την επιστημονική ε, θέση της επιστημονικής κοινότητα. Όπως ξέρετε, το πρόβλημα της θρησιμότητας των μελισσών είναι σύνθετο πρόβλημα, έχει πολλούς παράγοντες, πολλές αιτίες. Δεν είναι εύκολο να εντοπίσουμε με ακρίβεια ε, τα αίτια και, ω εκ τούτου είναι και πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο του φαινομένου αυτού. Και αυτό είναι ακριβώς ε, στην ίδια γραμμή με, και αυτό προκύπτει ακριβώς και από πολλές έρευνες που έχει χρηματοδοτήσει για το σκοπό αυτό η Επιτροπή και αυτό ήταν και το αποτέλεσμα της γνωμοδότησης που δόθηκε στην Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, την ΕΦΣΑ. Μετά από την άποψη της ΕΦΣΑ η Επιτροπή προσπαθεί να προχωρήσει σε μια σημαντική δραστηριότητα που είναι ο ορισμός ενός εργαστηρίου της Ένωσης, εργαστηρίου αναφοράς για θέματα υγείας μελισσών. Έχουμε μια μακρά εμπειρία στον τομέα των ευρωπαϊκών εργαστηρίων αναφοράς για την υγεία των ζώων, θετική σε μεγάλο βαθμό και θέλουμε να ε, χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία, αυτή και στον τομέα το, της μελισσοκομείας η διαδικασία ορισμού του εργαστηρίου αυτού συνεχίζονται. Το εργαστήριο θα είναι λειτουργικό ήδη κατά το πρώτο ήμιση του 2011 και θέλουμε να ξεκινήσουμε μαζί με τα εργαστήρια αναφορά σε ένα πιλωτικό σχέδιο εποπτείας της θνησιμότητα των μελισσών. Κάτι που, είναι σημαντικό, κάτι που είναι σημαντικό για να έχουμε εναρμονισμένα συστήματα εποπτείας που θα εξασφαλίζουν ασφαλή δεδομένα για το πρόβλημα. Διότι ένα από τα θέματα που σαφώς ανέκυψαν είναι και η έλλειψη ασφαλών στοιχείων για την, ε, τα χαρακτηριστικά του προβλήματος. Τα πιλωτικά λοιπόν σχέδια που προτίθεται να χρηματοδοτήσει η Επιτροπή και που τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενεργοποιήσουν είναι ακριβώς έχουν αυτό το στόχο, να καλύψουν το κενό αυτό. Ένα κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία των μελισσών είναι ε, εν πολύ συναρμονισμένο σε σχέση με μια σειρά ασθενειών εξωτικών και σε ό,τι αφορά την εσωτερική ε, τις εσωτερικές ασθένειες των μελισσών. Τούτο ισχύει και για τον έλεγχο των υπολοιμάτων στο μέλι. Υπάρχει ένα νομισμένο κοινοτικό πλαίσιο και έλεγχοι δημόσιας υγείας που εξασφαλίζουν ότι το εισαγόμενο μέλη από τρίτε χώρε στην Ένωση προσφέρει τις ίδιες υγειονομικέ εγγύησει με αυτό που παράγεται στην Ένωση. Μια σειρά... Ξεκινήσαμε επίση και μια σειρά δραστηριοτήτων στον τομέα των παρασυτοκτόνων. Η Επιτροπή βάση της δήλωσης που είχε υποβάλει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ξεκίνησε ήδη τι εργασίε αναθεώρηση των απαιτουμένων για την υποβολή των φακέλων παραστοκτώνων. Πρέπει να υπογραμμίσουμε επίσης ότι πρόσφατα χρηματοδοτήθηκαν για την επόμενη τριετία μια σειρά προγραμμάτων κρατών μελών υποστήριξης του κλάδου της μελισσοκομείας που συμπεριλαμβάνουν και δράσεις ελέγχου της τις ε, κάτι που είναι ε, σημαντικότερο, που αυξη, ποσοστό αυξημένο κατά 60% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η Επιτροπή Πρόεδρε θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μία ανακοίνωση σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της υγείας των μελισσών πριν τελειώσει το 2010, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ε, η Επιτροπή θα μπορέσει να έχει μια θέση όλων των ενδιαφερμένων πλευρών, ιδίω των ευρωπαϊκών θεσμικών προγραμμάτων, για το ζήτημα αυτό. Σα ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση. Το λόγο έχει πρώτα πρώτα η κυρία Λούλινγκ. Ε, ε, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστώ για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της και πάνω από όλα που υιοθέτησε ευθύς αμέσως στην πρωτοβουλία μου για μια συζήτηση ε, προφορική ερώτηση με συζήτηση και ψήφισμα διότι δυστυχώς ακόμη εφέτος δεν μπορούμε να κάνουμε έκθεση καθώς δεν έχουμε πλέον ε, πόντους ε, για να κάνουμε έκθεση για, την, για τον κανονισμό μάλλον του Συμβουλίου της 28 Μαΐου του 2010 για την εφαρμογή της ε, των μέτρων που ισχύουν για τα προϊόντα γεωργίας. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε λοιπόν, να συστήσουμε και πάνω απ' όλα να ευαισθητοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ώψη της ε, ε, ανακοίνωσής της ως προς το μέλλον της ε, ε κοινή γεωργική πολιτικής από το 2013 ε, και μετά. Θέλουμε εγκαίρως να ευαισθητοποιήσουμε λοιπόν την Επιτροπή και θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη αισθάνομαι προ του εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα ενημέρωσαν για τα όσα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε σχέση με προηγούμενε διεκδικήσει έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνουν πράγματα που έχουν ήδη γίνει, να μην διεκδικούμε πράγματα που ήδη έχουν γίνει μέσα στο ψήφισμα. Ευχαριστώ επίση όλε τι ε, πολιτικέ ομάδε που συνέβαλαν στην διατύπωση αυτή τη ε, προτάσεως ψηφίσματος που θα υποβληθεί στο δικό σας όνομα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εγώ να πω πάντως ότι κρίνω απολύτως ε, σημαντικό να πούμε αυτό που θεωρούμε ε, ότι πρέπει να είναι η εφαρμογή των μέτρων του κανονισμού που ισχύει το 1997 και να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι τα προγράμματα ενισχύσεων για την ε, ε, μελισσοκομεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η διάρκεια και η ουσιαστική τους, η αποτελεσματικότητά τους πάνω απ' όλα. Καλά είναι τα προγράμματα, αλλά το, βαθμός Εκτέλεσή τους ε, ποικίλει και ανάλογα με το κράτος μέλος αλλά και ανάλογα με το έτος εφαρμογής. Πρόσφατα στην Ιταλία σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, εκδήλωση για την εβδομάδα του μελιού στο Μονταλτσίνο που επισκέφθην Έμαθα ότι, και μάλιστα από την ίδια την εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι χρειάζονται καλύτερε στατιστικέ στη και μόνο 5 με 6 κράτη από τα 27 αξιοποιούν πλήρω τον προπολογισμό που έχουν στη θέσή του. Αν και η κατάσταση είναι βελτιούμενη και υπάρχουν πολλά και δεν υπάρχουν πλέον κράτη-μέλη που αξιοποιούν μόνο το 1 τρίτο των κονδυλίων όπως είχαμε δει το 2007. Το 2008, 2009, 12 ήταν τα κράτη που ξεπέρασαν το 80%, μάλλον 90% στην εκτέλεση και 7 εκείνα που έφτασαν στην εκτέλεση 100%. Θα ήθελα επίσης να πω δύο λόγια ως προς την εξέλιξη του αριθμού των μέλισσοκόμων και των κυψελών στα κράτη-μέλη. Στατιστικές για τα έτη 2003 και τις περιόδους 2004, 2008, 2010 είναι μάλλον αξιοπερίεργες για ορισμένα κράτη και διαρωτώ με κατά πόσο αυτές οι στατιστικές μπορούν να κρυθούν αξιόπιστες. Διότι ο προπολογισμό που έχουμε στη διάθεσή μας κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών επί τη βάση του αριθμού των κυψελών που έχουν. Διαπιστώνω λοιπόν, επί παραδείγματι, ότι για την Πολωνία, με βάση αυτές τις στατιστικές, οι μελισσοκόμοι από 42.800 έχουν γίνει 39.000. ενώ οι κυψέλες από 941.000 έχουν αυξηθεί στο 1.123.000. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς είναι δυνατόν ύστερα από μια ε, ε, αναδιάρθρωση τομέα να έχουμε τέτοιε αυξήσεις στις, ε, και, και, κυψέλες και αντίστροφα μείωση αριθμού μελισσοκόμων. Από την άλλη έχουμε κάποια εικόνα διαφορετική ε, εικόνα στις ε, επιμέρους περιφέρειες ως προς τον αριθμό αλλά και την ηλικία των μελισσοκόμων και μάλιστα των μη επαγγελματιών ε, μελισσοκόμων, των αραστεχνών μελισσοκόμων. Γι' αυτό θα ήταν καλό να αναπτύξουμε προγράμματα κατάρτισης ενημέρωσης των μελισσοκόμων, επαγγελματιών και μη και επισκοπεύω να κάνω μια σχετική τροπολογία στο σχέδιο της, του ψηφίσματος. Για τα φυτογεινά προϊόντα θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία και του συντονισμού πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ε, επισήμανσης ετικετοθεσίας δηλαδή για ορισμένα επικίνδυνα προϊόντα έτσι ώστε να έχουμε μέτρα περιορισμού των κινδύνων στα προϊόντα αυτά και έτσι ώστε να ισχύουν τα προγράμματα για ε, παρακολούθηση και έλεγχο της χρήσης φυτογεινών προϊόντων στις μέλισσες για να υπάρχει και η συγκρισιμότητα και βεβαίως ακούσαμε ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα εν εξελίξη στην υπόθεση αυτή κυρίως με το σχέδιο το πιλωτικό σχέδιο για το οποίο ανέφερε μόλι ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Ένα άλλο σημείο το οποίο επίση με ενδιαφέρει πολύ είναι αυτό των ζωονόσων που πλήττουν τις ε, μέλισσες και που πιστεύω θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν σε επίπεδο την ιατρικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 32 εκατομμύρια περίπου θα έχουμε στη διάθεσή μας για το επόμενο έτος, που όμως είναι ψίχουλα σε σχέση με την τεράστια σημασία που έχει η ε, μέλισσα για την επικονίαση στη φύση. Η δεύτερη ιατρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται να είναι σχεδιασμένη μόνο για ε, οι άσημες ε, νόσους ή ζωονόσους όμως δεν θα πρέπει τα, προγράμματα που χρηματοδοτούμε με τα ελάχιστα αυτά κονδύλια που έχουμε στη θέσή μας να πηγαίνουν μόνο σε τέτοιου είδους ε, μέτρα για το μέλι και τα προϊόντα του, αλλά θα πρέπει να τα αφιερώνουμε για κάθε είδου τρόπο προαγωγή μελισσοκομεία και όχι μόνο για τη μετώπιση των ζωονόσων. Υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία δηλαδή απορροφούν πολύ μεγάλο μερίδιο αυτών των κονδυλίων, κυρίω για την καταπολέμηση βαροάση, την οποία ε, είχαν καταπολεμήσει στο παρελθόν, χωρί όμω κοινοτική συμμετοχή. Τώρα απλώ του έρχεται πιο φθηνά αυτή η προσπάθεια, γιατί συμμετέχει κατά 50% στην χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ένωση μάλλον, και μέχρι τότε, τουλάχιστον δική μου η πατρίδα, ε, αναλάμβανε 100% τα έξοδα καταπολέμηση βαροάσει. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα θέλαμε να επιμείνουμε και να πείσουμε την Επιτροπή αυτέ τι επιζωονώσει να τι αντιμετωπίσει μέσα από την κτηνιατρική πολιτική και όχι μέσα από τη γεωργία. Είδαμε μάλιστα τα τελευταία χρόνια ε, σημαντική βελτίωση της παραγωγής και χάρη στην ε, ε, σημαντική εξέλιξη τα τελευταία περίπου 10 χρόνια της μοριακής βιολογίας ίσως το κοινό να μην έχει μπορέσει να παρακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις και να μην είναι ενήμερο ίσως και να αισθάνεται δέος εναντί αυτών των εξελίξεων που δεν μπορεί να αντιληφθεί είναι κατανοητό το να φοβάται κανείς αυτό που δεν γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει δεν πιστεύω όμως ότι θα πρέπει εμείς μέσα από το ψήφισμα για τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς να είμαστε τόσο τόσο πια επίμονη στην αναφορά σε αυτού. Ναι, μπορούμε να του επισημάνουμε, αλλά πρόκειται για έναν αγώνα, πιστεύω, τον οποίο θα πρέπει η Επιτροπή Αρμόδια για το Περιβάλλον ε, να αποδειθεί μαζί με του ειδικού, ε, του περιβαλλοντολόγου και όχι εμεί. Γιατί ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιο σχετισμό μεταξύ τη θνησιμότητα των μελισσών και τη χρήση κάποιων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, πλην όμω, σε φυτά, πλην όμω δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο μέχρι τώρα και οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στην Ευρώπη έχουν πολύ περιορισμένη καλλιέργεια. Είναι πολύ περιορισμένες οι ποσότητε δηλαδή καλλιεργουμένων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Και γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ορίσουμε και μια προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών, ώστε να είμαστε έτοιμοι, να τις λάβουμε όλες υπόψη και να κρίνουμε το πώς θα προχωρήσουμε στην ικανοποίηση των ετοιμάτων εκείνων των συναδέλφων που θα ήθελαν ακόμη να συμμετάσχουν στην επεξεργασία του ψηφίσματος. Κύριος όμως στόχος νομίζω θα πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για την διαφύλαξη, την συνέχιση καλύτερα και την ενίσχυση των μέτρων για την υποστήριξη της μελισσοκομίας και μέσα από τη νέα κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013 ήθελα δεν να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την συνεργασία εκ μέρου όλων ημών και να εκφράσω την ευχή πως θα καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα που θα ικανοποιεί τους στόχου και τους δικού μα και αυτού των μελισσοκόμων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λούλη. Κυρία Μορβάη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι με έχουν κατακλείσει οι Ούγγροι με με πλειάδα επιστολών όπου καταγγέλουν την, ε, τους κινδύνους και τις μεγάλες καταστροφές που τους απειλούν λόγω της πλεονεξίας ορισμένων κερδοσκόπων. Το παραδοσιακά καλό ουγγρικό μέλι κινδυνεύει. Κινδυνεύει η επιβίωσή του, κάτι το οποίο βλέπουμε όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά και σε άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται ε, μέλι παραποιημένο, μέλι που δεν είναι καθαρό και επίσης η πλεονεξία αυτών των κερδοσκόπων οδήγησε σε μόνο καλλιέργειες, σε μεγάλες εκτάσεις μόνο καλλιέργειας, στις οποίες και περιορίζεται βιοπικιλότητα αλλά και χρησιμοποιούνται ε, ζεσανιοκτώνα πολύ επικίνδυνα για, τα, για τη μέλισσα και την υγεία της. Ε, μεγάλο επίσης ε, πρόβλημα επισημαίνεται στο ότι οι διαφορετικές ε, μέλη διαφορετικών προελεύσεων και ποιοτήτων ε, αναμειγνύεται και φτάνει τελικά στον καταναλωτή με τη μορφή του μείγματος. Το πολύ γνωστό λοιπόν και διάσημο ουγγρικό μέλι, διάσημο για την φήμη του, για την ποιότητά του και γνωστό ανά τον κόσμο ουγγρικό μέλι, φαίνεται ότι φτάνει τελικά ε, μέσα σε ένα βάζο το οποίο περιέχει πολλά άλλα είδη μελιού, κινέζικο μέλι το οποίο κάκιστης ποιότητας ε, επιλέγουν οι κερδοσκόποι να ε, αναμίξουν με το καλό ουκρικό μέλι για να κερδίσουν όσο δυνατόν περισσότερο. Πράγμα το οποίο βεβαίως πλήττει βαθύτα, βαρύτατα και την φήμη του ουκρικού μελιού. Αλλά μάλλον αυτό το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην Ουγγαρία και το μέλι της. Παρακαλώ λοιπόν να ληφθεί υπόψη και το αίτημα των ε, Ούγγρων μελισσοκόμων για τον περιορισμό των ε, για την απαγόρευση της ανάμειξης αλλοδαπών προελεύσεων μελιού μέσα σε ευρωπαϊκό μέλι. Αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω ότι η καλή ε, τικητοθεσία, η καλή σήμανση θα έλυνε κάθε πρόβλημα. Θα έβλεπε ο καταναλωτής τι μέλι έχει το βάζο που σκοπεύει να αγοράσει και θα αποφάσιζε με βάση τα δικά του κριτήρια τι είδους μέλι θέλει να καταναλώσει. Γιατί βέβαια κάθε μελισσοκόμος, κάθε κυψέλη και κάθε κράτος ή περιοχή παράγει διαφορετικής ποιότητας και γεύση μέλι. Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό που έχει να κάνει με, τα, ε, με την ε, μη τήρηση ή ελλειπή τήρηση η, την απουσία ακόμη και ισχύω των μέτρων ποιότητας, ε, των προδιαγραφών ποιότητας που έχουμε για τα δικά μας προϊόντα στα προϊόντα που έρχονται από τα τρίτα κράτη. Πράγμα το οποίο έχει σαν συνέπεια τα ε, τρίτα αυτά κράτη να κατακλείσουν την ευρωπαϊκή αγορά με τα κακής ποιότητας, με τα κατώτερη ποιότητας αλλά και φθηνότερα δικά του προϊόντα. Αυτό που έχουμε πάθει δηλαδή εμεί στην Ουγγαρία με το μέλι. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορούσε ο Μελισσοκόμο και να απολύει το μέλη του στην περιοχή στην οποία είναι εγκατεστημένος, αλλά και ταυτόχρονα να συμμετάσχει μέσα σε ένα δίκτυο ε, εμπορία του μελιού ε, πιο οργανωμένο που θα το επέτρεπε με άμεση επικοινωνία με τον καταναλωτή, να διαθέτει το προϊόν αυτό και πιο μακριά από τη στενή του περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τραβήξουμε το χαλί κάτω από τα πόδια αυτών των μεγάλων διεθνών κερδοσκόπων που κάνουν τόσο κακό στους Ούγκρους ε, μέλισσοπαραγωγούς, με, ε, μελισσοκόμους. Και καλό θα ήταν να επανέλθουμε στο τι σημαίνει καλό και γνήσιο μέλι. Εμείς βλέπουμε να καταθέσουμε τροπολογίες μέσα στις ε, ε, προθεσμίες που έχουν οριστεί. Είναι καλό εν γέννη το κείμενο, όπω θα να κάνουμε μικρές βελτιώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη Ευχαριστώ. Η προστασία της σας ε, είναι ένας από τους κύριους στόχους που πρέπει να εξυπηρετεί η γεωργία, γιατί η μέλισσα και προστατεύει τη βιοπικιλότητα και εξασφαλίζει την επικονίαση και αποτελεί δίκτυο υγεία τη φύση. Έτσι λοιπόν, η μεγάλη χρησιμότητα ή ο περιορισμό ε, ε, του επαγγέλματο, η περιστολή του επαγγέλματο του μελισσοκόμου αποτελεί ένα κακό δείγμα ε, για τον τομέα τη μασολοκομία στην Ευρώπη που χρειάζεται κατεπηγόντω υποστήριξη. Υπάρχουν διάφορα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία τη μέλισσα. Θα μπορούσαμε όμω στο ψήφισμα αυτό να επικεντρωθούμε σε ορισμένα κεντρικά ζητήματα, όπω παράδειγμα τη συνέχιση των υφισταμένων προγραμμάτων για τις ε, μέλησες μέσα στις προσεχείς δημοσιονομικές ε, το δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2020. 20 επίσης ε, έρευνα ιδιαίτερα για το ρόλο της μεσλησοκομεία στη Γεωργία, όπου μπορούμε πολλά ακόμη να διδαχθούμε. Καλύτερη καταπολέμηση των επιζωτιών και των νοσογόνων παραγόντων, ιδιαίτερα της βαροάσης. Και

πιο ομοιόμορφε στατιστικέ στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση από όλα τα κράτη-μέλη, έτσι να μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα τα αποθέματα τη σα, Έχουμε πάνω από 600.000 μελισσοκόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί όμω να έχουμε παρκή στοιχεία για να γνωρίσουμε τι είδου αποθέματα σε μέλη σα έχουμε. Και γι' αυτό θα ήταν καλό να έχουμε ένα είδο εργαστηρίου αναφορά πάνω στο οποίο να μπορούμε να παραπέμπουμε και να ελέγχουμε τα αποθέματα. Καλύτερη και περαιτέρω κατάρτιση των ε, μελισσοκόμων, στην οποία θα πρέπει να επενδύσουμε και επίση θα πρέπει να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέου μελισσοκόμου έτσι ώστε να ενδιαφερθούν και να αναπτύξουν αυτή τη δραστηριότητα. Και επίσης θα ήθελα κλείνοντα να αναφερθώ σε ένα, σύντομο, σε ένα μικρό πρόβλημα ε, στη μετάφραση στο κείμενο του ψηφίσματος ε, βλέπω τη λέξη θνησιμότητα της σα, be mortality, ως ε, ε and sterben, ενώ θα έπρεπε να είναι and sterblichkeit, θνησιμότητα δηλαδή. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρσία Περές. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίηση για την πρωτοβουλία που λάβαμε ως Επιτροπή Γεωργίας. Είμαι βέβαιο ότι ο κλάδος της μελισσουργίας στην Ευρώπη θα υποδεχθεί θετικά την πρωτοβουλία αυτή, προφορική ερώτηση με ψήφισμα. Μιλάμε, Πρόεδρε, για ένα στρατηγικό κλάδο. Στρατηγικό γιατί υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της διαφύλαξης βιοποικιλότητας και της ενίσχυσης της ε, μελισσουργίας. Ε, είναι λοιπόν σημαντικός ο κλάδος αυτός για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ε, οι θέσεις που παρουσιάζονται στο ψήφισμα είναι θετικές για τον κλάδο, εκφράζει σωστά τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος, τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά του. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να τεθούν με μεγαλύτερη έμφαση. Έχουμε χρόνο για να υποβάλουμε τροπολογίες και να βελτιώσουμε το υφιστάμενο κείμενο. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε μέσω της εργασίας αυτής. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η μέλη σουργία εξαρτάται πολύ από τα εθνικά προγράμματα υποστήριξης που συχνά είναι ε, τα μόνα Επίσης, είναι σημαντικό να υπογράψουμε ότι το παράσιτο σκόρος βαρό δημιουργεί προβλήματα στην ε, μελισσοκομία, στη μικρή και μεσαία μελισσοκομία στην Ευρώπη. Πρέπει να δώσουμε έμφαση, έμφαση στην ανάγκη να βελτιώσουμε την, ε, υγι, την ποιότητα υγείας αλλά και τον έλεγχο στα κρατημέρια. Κατόπιν θα έχουμε χρόνο για να συμπεριλάβουμε και αυτά τα ζητήματα στο κείμενο του ψηφίσματος. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν που εξήγησε την κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει σε κάποιες αμφιβολίες που έχω ακόμα. Βλέπω ότι στο ψήφισμα αναφερθήκαμε στο ζήτημα της ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής κτηνιατρικής, ε, στην Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική ε, Επιτροπή και την ε, μελισουργία. Αυτό το ζητά ο κλάδος. Αλλά από όσο ξέρω υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κάποιες οργανώσεις του κλάδου που αμφισβητούν ή θεωρούν ότι δεν είναι θετική η συμπερίληψη του κλάδου στο, στην ευρωπαϊκή κτηνιατρική πολιτική. Ξέρει κάτι σχετικά η Επιτροπή. Θα μπορούσε να μου δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Γκαρσιαπερές, ο κύριος Νικολέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάβασα το σχέδιο ψηφίσματος και νομίζω ότι είναι ένα ψήφισμα που φτάνει στην κατάλληλη στιγμή και καλύπτει τα προβλήματα του μελισσοκομικού τομέα στην Ευρώπη. Έχω κάποιες προτάσεις να κάνω ωστόσο. Πρώτα απ' όλα, βεβαίω αναφέρεται το ψήφισμα στη σημασία των εθνικών προγραμμάτων για τη μελισσοκομεία για το έτος 2012. Όμως πιστεύω ότι θα έπρεπε να ζητήσουμε τα προγράμματα αυτά να εξακολουθήσουν και μετά το 2012. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναφέρουμε και τη ρήπανση. Ρήπανση η οποία πλήττει την μελισσοκομεία στην Ευρώπη. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που έλεγαν προηγουμένως ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε, να καλλιεργήσουμε την ανάπτυξη των τοπικών αγορών, ώστε να υπάρχει άμεσο συσχετισμό μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών. Αυτό θα είναι ευεργετικό και ωφέλιμο για όλα τα κράτη-μέλη και για την Ένωση γενικότερα. Έπειτα, θέλω να τοποθετηθώ κατά της πρωτοβουλίας να υπάρχει ένα σύστημα επιθεωρήσεων και ελέγχων για την υγεία των μελισσών. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά, αρκετούς τέτοιους οργανισμούς και φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, η πτυχή αυτή Ίσως δεν βρίσκει τη θέση της επαρκώς στο ψήφισμα αυτό και στο κείμενό μας, όμως θα έπρεπε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στους νέους μελισσοκόμους. Αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστίε προς την κυρία Λούλιν για το διαρκές ενδιαφέρον της για αυτό το τομέα. Η ψηφοφορία ε, για τον προπολογισμό στήριξε την αύξηση του κονδυλίου που προτείνεται για το χρόνου. Οπότε υπάρχει διαρκή στήριξη και από μας. Τώρα, κάποια σχόλια για το ψήφισμα. Εδώ υπάρχουν δύο τομείς αλληλένδετοι που πρέπει να εξετάσουμε παράλληλα. Η επαγγελματική μελισσοκομεία αλλά και η ιδιοπικιλότητα, για την οποία υπεύθυνη είναι και η μελισσοκόμη. Η παράγραφος 12 είναι πολύ σημαντική για τη μεταφορά γνώσης και την έρευνα από αυτούς που διαχειρίζονται το γεωργικό τοπίο και οικοτόπους, τοποθεσίες που μπορούν να ευνοήσουν την ε, διαβίωση των αγριομελισσών. Διότι με τη μελλοντική μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ θα πρέπει να προβλέψουμε αρκετή ευελιξία για τα κράτη-μέλη ώστε να εξετάσουν ενδεχόμενους τρόπους ενθάρρυνσης των γεωργών να εγκαθίστανται σε συγκεκριμένες περιοχές. Λόγου χάρη, δύο εκτάρια εκμετάλλευση ε, που άρχισε να λειτουργεί την περασμένη περίοδο, ε, την περασμένη σεζόν, ε, πέτυχε αρκετά, αλλά χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται κονδύλια για να πετύχει και έναν ικανό μελισσοκόμο. Ω προ του νέου μελισσοκόμου, συμφωνώ ιδιαίτερω, διότι δεν ενθαρρύνουμε επαρκώ του νέου να αφοσιωθούν σε αυτό το τομέα. Χρειάζεται ιδιαίτερη υπομονή και βαθιά γνώση και επιμονή για να πετύχει κανεί εδώ. Στηρίζω λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία και σε ό,τι αφορά τι βιοτεχνολογίε. Να πω ότι από του αριθμού που μα έχει δώσει η Επιτροπή η Κίνα, η Βραζιλία και οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι οι πρώτε στη χρήση βιολογικών τεχνολογιών. Εάν πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει συσχετισμό μεταξύ τη μείωση του πληθυσμού των μελισσών και τη χρήση των βιοτεχνολογιών, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα. Όμω δεν είμαστε βέβαιοι εάν ισχύει αυτό, γιατί δεν έχουμε τόσε πολλέ καλλιέργειε γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών στην Ευρώπη και εδώ έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού. Άρα Υπάρχει περιθέριο, περιθώριο εξέλιξης εδώ και στηρίζω την προσέγγιση της κυρίας Λούλιν σε αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε κυρία Μακίνες, ο κύριος Εκχάουτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη δουλειά σας για το ψήφισμα αυτό και την κυρία Λούλιν επίσης για το τόσο συστηματικό της έργο. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν και συμφωνούν το τι σημασία έχει ο τομέας της μελισσοκομεία για τη βιοπικιλότητα και την γεωργία γενικότερα. Νομίζω το πλέον σημαντικό για το συγκεκριμένο ψήφισμα, διότι με χαρά την Επιτροπή να δηλώνω ότι θα δημοσιεύσει η ανακοίνωση στο τέλος της χρονιάς, αλλά αυτό που θα περιέχει η ανακοίνωση είναι και αυτό που βασικά μας απασχολεί. Δηλαδή, ζωτική σημασία είναι να εξετάζουμε του διαφορετικούς παράγοντε. Εδώ μιλάμε ένα πρόβλημα, ένα τομέα στον οποίο ασκούνται πιέσει από διαφορετικέ ε, πηγέ. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε τι κατάλληλε ε, λύσει για την κάθε περίπτωση και θα πρέπει το ψήφισμα να φέρει του διαφορετικού αυτού παράγοντε. Κάποιοι δεν αναφέρουν καν τι βιοτεχνολογίε, δηλαδή του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού. Ίσως να υπάρχει συσχετισμό, μα λένε οι επιστήμονε. Άρα αυτό που πρέπει εδώ να μα απασχολήσει είναι ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα και μάλιστα ανεξάρτητη. Πρέπει να είναι αξιόπιστα τα δεδομένα που ε, θα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν πολλέ επιτόπιε έρευνε, αλλά δεν είναι διαθέσιμε οι πληροφορίε. Να τι πρέπει να μα ε, απασχολήσει λοιπόν. Να ζητήσουμε από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή τη να αναφερθεί στο ρόλο των ε, παραστοκτώνων αλλά και των γενετικών τροποποιημένων οργανισμών όλων των παραγόντων που ε, ε, αναφέρονται στο ψήφισμα. Να ζητήσουμε έρευνα όμως, περαιτέρω μελέτες, ώστε να διατεθούν δημοσίως και αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να ζητά το ψήφισμα. Είναι πολύ ευγενή ο σκοπό μα και πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτή τη γραμμή. Για να είμαστε βέβαιοι ότι η έρευνά μα θα συλλέγει τέτοιου δεδομένα. Και εν τέλει να γνωρίζουμε ποιοι παράγοντε πραγματικά επηρεάζουν. Η κυρία Μαγκίνε, ναι, υπάρχουν μέλησης και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά και αλλού υπάρχουν προβλήματα και στην Αμερική μάλιστα τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα και εκεί χρησιμοποιούν και περισσότερο του γενικού τροποποιημένους οργανισμούς. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν συσχετισμό, απαιτείται έρευνα και αυτό ακριβώ ζητά το ψήφισμά μα. Ε, ε, προσδοκώ λοιπόν ότι ω Ευρωκοινοβούλιο θα ζητήσουμε τέτοιου είδου έρευνα και θα ακολουθήσουμε πιστά αυτή τη γραμμή, όπω αναφέρεται και στο ψήφισμά μα. Ευχαριστώ, Γκλάτενφελντερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα να επισημάνω, να σας αναφέρω μια ιστορία. Το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε η μητέρα μου ήταν ένα, μια σχολή μελισσοκομείας για πολλά χρόνια. Ε, πριν ε, να γεννηθεί η μάνα μου, το οποίο όμως ε, κατέλαβαν οι κομμουνιστές, το κρατικοποίησαν και το διάθεσαν για κατοικία. Για κατοικία. Δεν είχαν φυσικά λόγο σε αυτή την υπόθεση με λησοκόμη, όπω και δεν έχουν και τώρα με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θέλω να πω ότι αυτό το ψήφισμα έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, ότι δηλαδή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει μετά το 2013 και στο πλαίσιο τη κοινή γεωργική πολιτική να εξασφαλίσει την. να ενισχύσει τις ενισχύσεις που χρειάζονται, την υποστήριξη που χρειάζονται οι μελισσοκόμοι Θα ήθελα επίση να επισημάνω, για να συμπληρώσω την πρόταση, ότι στο επόμενο εξάμεινο, όπως μας ανέφερε χθε ο επίτροπο, Τσόλο, θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία πρόταση για την πολιτική ελέγχου της ποιότητας στα γεωργικά προϊόντα. Θα ήταν καλό λοιπόν να, ασχοληθούμε και να ασχοληθεί και με τη μελοσοκομεία στο πλαίσιο αυτή τη ε, πρωτοβουλία. Καλό θα είναι να έχουμε μια ικανοποιητική επισήμανση στα προϊόντα ε, του μελιού που έρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Γιατί αν αγοράσω ένα βάζο ε, μέλι το οποίο περιέχει κατά 99% μέλι Αργεντινής και μόνο 1% μέλι ευρωπαϊκό, θέλω να πουθενά αυτό το ποσοστό, δεν αναφέρεται το 90% μέλη από την Αργεντινή και 1% ευρωπαϊκό μέλη, αναφέρεται μόνο ότι είναι μείγμα μελιών, τίποτε άλλο όμως. Ως εκ τούτου η ε, προστασία του καταναλωτή δεν εξασφαλίζεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό για λόγους ακριβώς προστασίας του καταναλωτή να είναι σαφές, ε, σαφής η αναγραφή πάνω στην ετικέτα του ποσοστού της προέλευσης ε, του κάθε είδους μελιού που μπαίνει μέσα στο βάζο. Επίσης θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε τον έλεγχο της αναφοράς σε μία ετικέτα προϊόντων που υποτίθεται ότι περιέχουν μέλι γιατί βλέπουμε στις συσκευασίες διάφορων προϊόντων ε, αναφορές ή εικόνες που μας παραπέμπουν στην ε, περιεκτικότητα σε μέλη. Εάν όμως κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, βλέπουμε ότι το προϊόν αυτό έχει μόνο 5% μέλι και, μόνο, και κατά 95% ζάχαρη. Εάν λοιπόν πρόκειται για προϊόν το οποίο δεν έχει επαρκή ποσοστά μελιού και έχει μόνο 5% μέλι περιεκτικότητα, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίζουμε ως προϊόν μελιού. Πρέπει να έχει διαφορετική περιγραφή στην ετικέτα. Είναι πιστεύω αυτό ένα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να εγκύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσκύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, πρότασή της. Αυτό εν γέννη και για άλλα προϊόντα και εν γέννη στο ε, τομέα της πολιτικής επαλήθευσης και προστασίας της ποιότητας των προϊόντων μας. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε την συζήτηση με τον συνάδελφο. Σύντομα, για το θέμα των μελισσών, ο ρόλος της αλυσίδα βιοπικιλότητας και ο ρόλος του στη βελτίωση της βιοικής παραγωγής είναι αδιαμφισβήτητος πλέον. Αντίθετα, και το είδαμε αυτό στη συζήτηση, τα αίτια της θνησιμότητάς τους αποτελεί αντικείμενο θερμής συζήτησης. Άλλοι, κάποιοι δηλώνουν ότι φταίει αυτό με εξαιρετικό ενθουσιασμό, άλλοι εξηγούν ότι το ανάπορο ακριβώς οδηγεί σε θνησιμότητα των μελισσών. Νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει πραγματική δουλειά στην ε, ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων για την αναζήτηση των πραγματικών αιτιών της θνησιμότητας των μελισσών, να το βγάλουμε από την πολιτική συζήτηση και να το κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Διότι επαναλαμβάνω ότι η μέλισσα δεν έχει μόνο ρόλο παραγωγής μελιού, αλλά και καλής λειτουργίας της βιοπικιλότητας. Ευχαριστώ. Για να κλείσει τη συζήτηση θα δώσω τον ε, ρόλο στον ε, Λαντομάντα, στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ο κ. Λαντομάντα έχει το λόγο να απαντήσει. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πήραμε και άλλα στοιχεία περαιτέρω μελέτης ε, ως Επιτροπή για μια σειρά πολύ σημαντικών ζητημάτων. Προσωπικά έλαβα κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις τις οποίες μπορώ να απαντήσω νομίζω. Ιδίως σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τις ε, νόσους, τις ε, των μελισσών. Τέσσερις υπάρχουν αυτή τη στιγμή που θεωρούνται μείζον σημασία σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής. Η πανόλη, η ευρωπαϊκή πανόλη, η αμερικανική πανόλη, το παράσιτο small eye beetle και η τρόπιλελαψ. Αυτές οι τέσσερις ε, μολυσματικές αιτίες είναι ε, οι βασικές αιτίες θανάτου των ε, ε, μελισσών και υφίστανται νομοθετική αντιμετώπιση. Εμάς μας ανησυχεί ιδιαίτερα το θέμα των εισαγωγών της εισόδου δύο παρασίτων, της τροπιλέλαψ και του small eye beetle που μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε απόλυτη προστασία στα σύνορα της Ένωσης για τέτοια παράσιτα, διότι μπορούν να εισέλθουν στο έδαφος της Ένωσης μέσω μια σειρά ε, φυτικών και μη φυτικών ακόμα προϊόντων που αναπόφευκτα ε, μπαίνουν στην Ένωση. Άρα υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος που δεν μπορεί να μηδενιστεί. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε το κοινοτικό πλαίσιο δεν επιβάλλει συγκεκριμένους κανόνες ε, για την, ε, τον, ε, το, το σκόλικα βαρόα που είναι πλέον ένα παράσιτο διαδεδομένο σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Άρα το να επιβάλλουμε κανόνες στο εσωτερικό της Ένωσης σημαίνει ότι θα δημιουργούσαμε απλά και μόνο περαιτέρω προβλήματα στους μελισσοργούς. Όπως είπα ωστόσο νωρίτερα και όπως κάποια μέλη της Επιτροπής υπογράμμισαν ήδη, χρήμα, συγχρηματοδοτούμε σαν Επιτροπή εθνικά προγράμματα που έχουν στόχο την καταπολέμηση της ασθένειας αυτής. Από την άποψη αυτή λοιπόν και εδώ είμαστε δραστήριοι. Το τι θα γίνει στο μέλλον. Η Επιτροπή σχεδιάζει μία πρόταση για ένα νέο νομοθετικό κείμενο υγείας των ζώων, έτσι ας το αποκαλέσουμε, ε, που θα καλύπτει όλα τα ζωικά είδη και τις μέλισσες βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κομισιόν ή η Ένωση θα πρέπει να ασχολείται με την υγεία των βατράχων, αλλά των... Αλλά η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να είναι μια προσέγγιση που θα καλύπτει σημαντικά είδη που θα, τύχει, που θα πρέπει να τύχει και, την υποστήριξη του Κοινοβουλίου που σχολίασε και την σχετική ε, ανακοίνωση, θα σχολιάσει και τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής. Το μέλλον της ανακοίνωσης, η ανακοίνωση που ετοιμάζουμε και που θα εγκριθεί μ, κατά πάση πιθανότητα πριν το τέλος του έτους, έχει στόχο κυρίως να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγεία των μελισσών. Σε ό,τι αφορά του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, όπω γνωρίζετε, η το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει να χορηγούνται άδεια καλλιέργεια μετά τέτοιων προϊόντων, μετά από ειδική άδεια ασφάλεια τη ΕΦΣΑ, που περιλαμβάνει και την εξέταση των διαστάσεων πιθανών συνεπειών αρνητικών συνεπειών των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, και στις μέλισσες. Όπως είπε και κάποιος άλλος βουλευτής, δεν υπάρχει ακόμα απόδειξη ότι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στην υγεία των μελισσών σε σχέση με μη τροποποιημένους γενετικά οργανισμούς. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Σας θυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 6η Οκτωβρίου και η έγκριση στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 26-27 Οκτωβρίου. Η κυρία Λούλιν έχει ξαναζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους και τα σχόλιά τους. Πολύ θετική συνεισφορά. Να πω τον Ούγκρο συνάδελφο ότι ασχολούμαστε εδώ και 10-15 χρόνια περίπου, για να μην πω παραπάνω, με την ετικετοθεσία. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε περαιτέρω κι άλλο στο ψηφισμά μας στο σημείο αυτό. Εγώ έχω κάποια στατιστικά στοιχεία στα χέρια μου που λένε ότι η τιμή εισαγωγή του μελιού κυμαίνεται από 1,24 ευρώ το κιλό Πράγμα αδύνατο. Δεν μπορεί να γίνει καλό μέλι με τέτοια τιμή. Και φτάνει τα 4,5, τα 4,5 ευρώ το κιλό από τη Νέα Ζηλανδία, ας πούμε. Εγώ θα υποβάλω τροπολογίες για να επιμείνουμε περισσότερο στα προβλήματα της ετικετοθεσίας. Όμως πρέπει να πω ότι τα προγράμματα επιτρέπουν πολλά από αυτά που αναφέρθηκαν και να θυμίσω ότι πριν από χρόνια Είχαμε ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει συγχρηματοδότηση 75% των μέτρων στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού. Ποτέ δεν συμφωνήσαμε ωστόσο, γιατί αν σε ορισμένε περιοχές δεν χρησιμοποιηθούν ολόκληρα τα κονδύλια που διατίθενται, αυτό συμβαίνει γιατί οι περιοχές, οι περιφέρειες και τα κρατη μέλη δεν έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση. Εάν η Επιτροπή δεν κατανοήσει ότι μπορούμε να εξεύρουμε κάποια εκατομμύρια για να εξασφαλίσουμε την παραγωγή των οποροκυπευτικών μας και των δημητριακών μας, ε, ας πάψουμε εδώ να συζητούμε. Ο κύριος Μπαρόζο κατάφερε να βρει ένα δις εξέφνης μάλιστα για την αναπτυξιακή βοήθεια. Και δεν μπορούμε εμείς να βρούμε μερικά εκατομμυριάκια για να εξασφαλίσουμε τη διαβίωση αυτών, την επιβίωση αυτών των προγραμμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να εμπλουτίσουμε το ψήφισμα και θα ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις ε, συμβολές τους. Ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ, ευχαριστούμε και την Επιτροπή και όλους τους συναδέλφους και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πράσινη βίβλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προετοιμασία των δασών εν ώψη τη κλιματική αλλαγή. Το σημείο αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπως θα ξέρετε. Όμως θα πρέπει και εμείς να υποβάλουμε τη δική μας νομοδότηση. Η Ευρω... Εξ ονόματος της δικής μας λοιπόν Επιτροπής έχει αναλάβει ο συνάδελφος ο κ. Νικουλέσκου. Να σας πω ότι είναι πολύ σημαντική εδώ. Βαρύνει ιδιαίτερα η νομοδότηση της δική μα επιτροπή, γιατί το θέμα αυτό έχει προκαλέσει μεγάλες ε, ε, συγκρούσεις μεταξύ ημών και της Επιτροπής περιβάλλοντος. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα καθορίσουμε τη στάση μας. Μιλάμε για τα δάση και τη συνεισφορά τους στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες ε, ως δημοσιογαθό. Γι' αυτό λοιπόν δίνω αυτή στο αμέσως το λόγο στον συνάδελφο Νικουλέσκο για να μας παρουσιάσει την πρόταση αυτή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μεγάλο το θέμα. Δεν θα προσπαθήσω να το καλύψω πλήρως τώρα. Η πράσινη βίβλος περιλαμβάνει τα βασικά, περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών δασών και τα προβλήματα που υπάρχουν για όλα αυτά τα δάση. Επίσης θέτει μια σειρά ερωτημάτων για να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος. Είναι γεγονός ότι τα δάση παρέχουν διαφόρου τύπους υπηρεσίες. Η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει προφανώς το δάσος. Ταυτόχρονα επίσης πρέπει να διαπιστώσουμε ότι αλλάζουν, αλλάζει η πανίδα και η χλωρίδα στα ευρωπαϊκά ε, δάση λόγω και της αλλαγής ε, του κλίματος ε, που καθιστά ευπαθέστερα τα δάση. Η πράσινη βίβλος προσπαθεί να απαντήσει σε κάποια τέτοια ερωτήματα. Τι ρόλο παίζουν τα δάση στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Πρέπει να αυξηθεί ο ρόλο αυτό Και αν ναι, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και με ποιο τρόπο πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο αυτό. Πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει, ποιε είναι οι περιοχέ που είναι πιο ευάλωτε λόγω τη αλλαγή του κλίματο και ποιο είναι ο τρόπο που μπορεί να έχει η Ένωση για να συμβάλλει στην δράση που ήδη έχουν ε, ε ξεκινήσει τα κράτη-μέλη. Άλλη ερώτηση. Η ευρωπαϊκή και οι εθνικές ε, πολιτικές μέχρι τώρα είναι επαρκής, συμβάλλει επαρκώς η Ένωση στην προστασία του δάσους. Πώς μπορούμε να δράσουμε για να διαφυλάξουμε την ε, δασική γεννητική κληρονομιά. Και τέλος, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, πληροφορίες ε, για την κατάσταση των δασικών αποθεμάτων. Η Κομισιόν θέτει δύο άξονες συζήτησης. Πρώτον, προστασία των δασών από την εμπορική εκμετάλλευση. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να μιλήσουμε εδώ για μια καλύτερα για μια σωστή διαχείριση των, ε, του δασικού πλούτου, διότι το δάσος συμβάλλει στη γεωργία, συμβάλλει στην επίτευξη μια σειρά κοινωνικών ή περιβαλλοντικών στόχων. Ε, είναι μια σημαντική πηγή ε, εσόδων για τις κοινότητες αστικές και ε, αγροτικές. Η διαχείριση των δασών ε, συμβάλλει στην οικονομία της υπαίθρου. Παρέχει θέσεις εργασίες και προσφέρει λύσεις για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι λοιπόν το δάσος ένα δημόσιο αγαθό. Τη συζήτηση αυτή την είχαμε κάνει στα πλαίσια μιας ε, συζήτησης για το μέλλον της ΚΑΠ και θεωρώ ότι η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τους ε, ιδιοκτήτες των δασών με χρηματοδότηση, ε, ειδική χρηματοδότηση για να, μπορέσει να, να μπορέσουν να αντισταθμίσουν κάποιες ζημίες που αντιμετωπίζουν. Έτσι θα προστατεύσουμε και τη βιοπικιλότητα. Δεύτερος άξονας συζήτησης, η παρέμβαση της Ένωσης εδώ. Έχουμε δύο επιλογές. Να διαφυλάξουμε την δασική πολιτική ως αρμοδιότητα των κρατών μελών ή να μετατρέψουμε να έχουμε μια κοινοτική δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Δεδομένων των, του, του κατεμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωση και κρατών μελών στη συνθήκη και τη αρχή τη επικουρικότητα, δεν πιστεύω ότι πρέπει να επεκτείνουμε τι αρμοδιότητε τη Ένωση στον τομέα του, στο δασικό τομέα. Η Ένωση έχει ήδη ισχυρή εργαλεία για την προστασία των δασών. Υπάρχει για παράδειγμα το πρόγραμμα Natura 2000. Έχει και άλλα παρόμοια μέσα για να προστατεύσει τα δάση. Να υπενθυμίσω ταυτόχρονα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε πλιστάκης άποψη η θέση υπέρ πραγματικά δασικής πολιτικής που θα μπορεί να εξασφαλίσει μια βιώσιμη διαχείριση των δασών και θα αναδεικνύει την σημασία τους. Η βιώσιμη ανάπτυξη του δάσους πρέπει να διεξάγεται, να έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Ευρωπαίου πολίτη. Διότι τα αγαθά που μπορεί να προσφέρει το δάσος βελτιώνονται. Η, δασοπον, η δασοκομεία και η δασοπονία μπορούν να τύχουν λοιπόν να έχουν μια ευρωπαϊκή διάσταση και πέραν της ε, και η προστατευτική αυτή προσέγγιση είναι τεχνητή. Προφανώς πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της γεωργίας και της δασοπονίας. Αλλά αυτό θα γίνει με μια καλύτερη ε, κατανομή της, ε, των ευθυνών μεταξύ των μεν και των δε. Δεύτερον, υπάρχει ο δεύτερος ε, πυλώνας της, Ευρω... της ευρωπαϊκής κοινή γεωργικής πολιτικής που πρέπει να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί με τη διαμόρφωση ε, σχεδίων ανάπτυξη υπαίθρου και με το 2013. Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή δράση στον τομέα του, του δάσους, τι χρειάζεται να γίνει. Προφανώς η αλλαγή του κλίματος θα έχει διαφορετικές συνέπειες στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Τα ευρωπαϊκά δάση θα μπορούν, του, της Βόρειας Ευρώπης θα μπορεί να γίνουν πιο παραγωγικά, ενώ τα δάση του Νότου να επηρεαστούν περισσότερο. Κατόπιν, ο, η προσαρμογη βαθμός προσαρμογής των ειδών διαφέρει στις υπηρετικές περιοχές όπου υπάρχει ήπιο κλίμα αλλού η προσαρμογή των ζώων να είναι δυσχερέστερη. Να υπάρχουν ακραία φαινόμενα σε κάποιες περιοχές πιο συχνά. Επίσης μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα υπάρξει μείωση των δασών στην Νότια Ευρώπη και σημαντικές αλλαγές. Γι' αυτό η στρατηγική προσαρμογή θα πρέπει να αποφασίζεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να συντονίζεται σε ευρωπαϊκό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, πληροφορίες που σχετίζονται με τον τομέα του δάσους. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα νέο στατιστικό εργαλείο που να περιλαμβάνει σαφείς πληροφορίε για το, την κατάσταση της υγείας των δασών, τη διατήρησή τους, να περιλαμβάνει σαφείς δείκτες δεδομένων για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα δάση, καλύπτοντας έτσι όλες τις ε, διαστάσεις που έχουν να κάνουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη των δασών. Εν, εν τέλει θα πρέπει να υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες αναδάσωσης στην Ένωση και σε εθνικό και σε τοπικό. Ζητάμε τα έργα αυτά να μπορούν κατόπιν να χρηματοδοτηθούν και με το 2013. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Νικουλέσκο. Να ξεκινήσουμε αμέσως τη συζήτηση. Είναι πολύ. οι συμμετέχοντες. Μα αμέσως μετά θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Σούλτ. Ξεκινάμε με την κυρία Εκ. Χωρίς μικρόφωνο. Δεν το είχα ανάψει. Mm, καλύτερα τώρα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ την ε, τον Σιτή για το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα, η δεσκομία, πάρα πολύ σημαντικό ως ευρωπαϊκό θέμα. Καλύπτει μεγάλο ποστό των εκτάσεων της Ευρωπαϊκής Επικράτειας, 40% όμως που το έχουν συστήσει πάρα πολύ λίγο. μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το ότι τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν μία μακροπρόθεσμη και ε, ανωδική κάλυψη των ε, εκτάσεων μας με δάση, πράγμα το οποίο είναι βέβαια πολύ θετική εξέλιξη για λόγους σεβασμού και της βιοποικιλότητας, προσθέσει οικονομίας, ανάπτυξης, κοινωνικών ε, εξελίξεων, αλλά και για λόγους προστασίας του κλίματος. Σκιώδη συγκήτρια δεν είμαι μόνο εδώ εκ μέρου τη Άλντε, αλλά είμαι και η σε επίπεδο Επιτροπή Βιομηχανία για την έκθεση αυτή και θα ήθελα να σημειώσω και να υπογραμμίσω ότι ο τομέας αυτός έχει ένα κύκλο εργασιών πάνω από 280 δισεκατομμύρια ευρώ, τεράστιο ποσοστό δηλαδή του συνολικού ΑΕΠ και 350.000 επιχειρήσεις που στηρίζουν τις δραστηριότητες τους στην δασοκομεία ε, και 8,6% της συνολικής μεταποιητικής, ε, του συνολικού μεταποιητικού εργατικού δυναμικού έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα πολύ σημαντικό οικονομικό τομέα. Βιώσιμη διαχείριση των δασών αλλά και η προστασία των δασών είναι πολύ σημαντική και για την ε, διαφύλαξη της βιοποικιλότητας αλλά και για την ε, συγκράτηση διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Η καλύτερη μέχρι τώρα τουλάχιστον μέθοδος για συγκράτηση, για περιορισμό των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα είναι να κόβουμε τα δέντρα και να τα ε, φτιάχνουμε να τα κάνουμε σπίτια όλα αυτά τα χρόνια. Παλιά και αποδεδειγμένα καλή μέθοδος. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε την ε, δασοκομεία κατά τρόπο όμως ανταγωνιστικό. Όχι μη ανταγωνιστικό, όχι δηλαδή να χαθεί η ανταγωνιστικότητα της ε, δασοκομείας και της ξύλο ε, της κοπής των ξύλων ή της αξιοποίησης του ξύλου. Με συγχωρείτε μπορείτε να με σταματήσετε να μιλάτε, δεν ακούτε τι λέω. Να μην σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε δηλαδή, τα προϊόντα των δασών και αντί αυτά, αυτό να εισαγάγουμε πλαστικό ή άλλα σύνθετα προϊόντα. Και πρέπει να υπογραμμίσω στην αρχή τη συζητήσεω αυτή ότι εδώ έχουμε και ζητήματα ιδιοκτησία. Να κρίνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το κείμενο της Επιτροπής είναι καλό κατά βάση. Καλωσορίζω την πρωτοβουλία, χαιρετίζω τις προθέσεις που αναπτύσσονται στο κείμενο. Πρέπει όμως να είμαστε και βέβαιοι ότι οι πρωτοβουλίες για, το δάσος, για τα δάση θα ενισχύουν τις ε, ε, αλλαγές, εξελίξει δάση και όχι μόνο θα τα προστατεύουν. Βλέπουμε κάποιες αλλαγές, υπάρχουν ήδη που ανεβαίνουν προς το βορρά όπως και ήδη εντόμων που σιγά σιγά εμφανίζονται στον βορρά. Έχουμε ήδη σκαθαριών τα οποία ήδη αποτελούν πρόβλημα στον Καναδά και τώρα βλέπουμε να εισβάλλουν και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα προς τα, βορειά της. Ε, πρέπει να βελτιώσουμε και την ενημέρωση του κοινού για τα χαρακτηριστικά του δάσους, ε, τα πλεονεκτήματά του, τα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές, τη συγκράτηση του εξίδου του άνθρακα, τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των δασών και επίσης θεωρώ ότι ο προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών και προδιαγραφών, όπως είπε και ο εισηγητής και χαίρομαι για την επισήμανση αυτή, πρέπει να αποτελέσει έναν τρόπο για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μα για βελτίωση τη κατάσταση στα δάση. Πράγμα το οποίο ακόμα δεν έχει συζητηθεί επαρκώ σε διεθνέ επίπεδο. Επίση, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο υπάρχει σημαντικό βαθμό επικουρικότητα, ω εκ τούτου ευρωπαϊκέ πρωτεγραφές μπορούμε να έχουμε μεν, ευρωπαϊκέ κατευθυντήριε γραμμέ μπορούμε να έχουμε μεν, πάντα όμω μέσα στο σεβασμό τη επικουρικότητα. Τα δάση είναι σημαντικά και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Άρα πρέπει και σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής να εξεταστεί αυτή η πτυχή. Ενισχυμένη συνεργασία και προσπάθειε για καλύτερη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μεταξύ Ένωση και κρατών μελών, πιστεύω, θα συμβάλλουν τα μάλα στι εξελίξει αυτέ και στου επιδεκόμενου στόχου. Και συμφωνώ κλείνοντα με τον εισηγητή ότι ε, επικρατούν μεταξύ Βορρά, Νότου, Ανατολή, Δύση Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πολύ διαφορετικέ συνθήκε και ω προ τη διαχείριση και ω προ την ιδιοκτησία, ω προ τι παραδόσει, την ιστορία και βέβαια των κρατών αλλά και τη βιοπικιλότητα. πρέπει δεν να βρούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα, μια φόρμουλα που να επιτρέψει την ε, συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών δεδομένων. Γιατί βλέπουμε από την ε, από το ιστορικό της νομοθετικής παρέμβασης επί Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν την ε, διαχείριση των δασών, μάλλον όταν αναλαμβάνεται σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, χείριση των δασών, συνήθω χάνεται και η επιχειρηματικότητα και η θέση εργασία. Και πρέπει να έχουμε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Εκ και τώρα κυρία Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που το ζήτημα αυτό το συζητάμε σήμερα, διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό συνολικά και από περιβαλλοντικής άποψη και επειδή έχει άμεση επίδραση και στον γεωργικό τομέα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ε, παρουσίαση από τον εισηγητή μας, πρέπει να πω ότι μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η παρουσίασή του, η επισκόπησή του, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και προβληματικών θα απασχολήσουν το Κοινοβούλιο στην αποτίμηση του όλου ζητήματος. Να πω λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ ευρύ στο σύνολο των τομέων που καλύπτει. Η δασοκομεία θα πρέπει να ε, υιοθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση. Διότι αν το κάνουμε αυτό από τώρα δεν θα καταλήξουμε σε αποτελέσματα διαρκή. Είναι πάρα πολλέ οι συνιστώσει αυτού του θέματο. Πρέπει επίση να πω ότι θεωρώ ε, ότι εδώ ε, μπλέκεται ιδιαίτερα και η εθνική αρμοδιότητα. Υπάρχει ανάγκη συντονισμού και συνεργασία. Αυτό θα πρέπει να είναι η πρώτη μα προτεραιότητα. Νομίζω ότι το ζήτημα που σήμερα συζητούμε αποτελεί μια μελλοντική πρόκληση για τη συνεργασία μεταξύ κατομελών και το συντονισμό που θα οργανώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπ' αυτήν την έννοια θα πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να επιτρέψουμε σε θετικές δράσεις να αναπτυχθούν και να μειώσουμε το κόστος. Εδώ θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. Να δαπανίσουμε λιγότερα. Εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν, νομίζω ότι εδώ πρέπει να ακολουθήσουμε δύο βασικές γραμμές δράσης. Η μία να αφορά την ανάπτυξη προπαρασκευαστικών δράσεων για τα δάση, προκειμένου να μπορούν να υποστούν τις κλιματικές αλλαγές, άρα προσαρμογή των δασών και επ' αυτού του θέματο έχουμε μια τεράστια πρόκληση μπροστά μα, διότι ξέρουμε ότι τα δάση από μόνοι του αποτελούν μια αυταξία και έχουν χαρακτηριστικά και ανάγκε τόσο διαφορετικά στα διάφορα μέρη και περιοχέ τη Ευρώπη. Όμω εδώ υπάρχει και άλλη μια συνιστόσα που πρέπει να λάβουμε υπόψη, ένα σκέλο που δεν μπορούμε να παραμελήσουμε. Η προστασία δηλαδή. Όχι μόνο η προετοιμασία, αλλά και η προστασία των όσων ήδη έχουμε. Χρειαζόμαστε να προστατεύσουμε, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα δάση που ήδη υπάρχουν και παράλληλα να αναπτύξουμε δράσει προετοιμασία και προσαρμογή για τι επερχόμενε κλιματικέ αλλαγέ. Επιτρέψτε μου στο σκέλος της προστασίας να προσθέσω κάτι ακόμη, διότι νομίζω ότι αυτό είναι το σκέλος που μας απασχόλησε λιγότερο ω τώρα, να πω τα εξή ότι αυτή η στιγμή είναι μια από τις πιο ανησυχητικές, ιδίως Εάν εδώ αναφέρουμε εντυπωσιακά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα μου, την Πορτογαλία, στοιχεία που δείχνουν ότι φέτο οι βασικές πυρκαγιέ ε, στην Πορτογαλία φτάνουν το 75% των ε, εκτάσεων που συνολικά ε, επλήγησαν από πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε τι διαστάσεις έχει αυτό το φαινόμενο και καταλαβαίνετε πόσο το τομέα της δασοκομείας στην Πορτογαλία εκπροσωπεί το 13% του ΑΕΠ και απασχολεί 7.000 μας. Έτσι λοιπόν για την προστασία νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει την απαραίτητη προσοχή ο υφηγητής, καθώ και στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να αναπτύξουμε δράσει απλώ ε, με το μέλλον ως γνώμονά μας. Είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάσουμε τα δάση για τις κλιματικές αλλαγές, κανεί δεν το αρνείται, αλλά αν δεν προστατεύουμε αυτά που ήδη έχουμε στα χέρια μας, όχι μόνο την προστιθέμενη αξία του θα χάσουμε, αλλά αν καούν αυτά τα δάση, θα επιβαρυνθούν τα προβλήματά μας με τις κλιματικέ αλλαγέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία πατραουνέβε, ο κύριο Γκάταφελντερ az előadó nagyon Πρόεδρε, νομίζω ότι ο συγκητής επισήμανε κατά εξαίρετο τρόπο ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε όλο και μεγαλύτερε πιέσει ε, στα δάση τη Ευρωπαϊκή, ει βάρο των δασών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναζητήσουν λύσει που θα συμβάλλουν στην φύτευση ειδών δέντρων που είναι τα καταλληλότερα ανάλογα με την περιοχή, εκεί που μπορούν να ευδοκιμήσουν τα είδη ανάλογα με τις κλιματικές και γεωφυσικές συνθήκες. Ίσως δεν θα έπρεπε να αναλογιστούμε και την απαγόρευση ε, φύτευσης ειδών δέντρων που δεν είναι ε, αυτοφυή σε μια περιοχή. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι θα ήταν σκόπιμο όταν ε, έρχεται η ώρα να συζητήσουμε τα θέματα αυτά της δοσοκομείας να επαληθεύουμε όλο το θέμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Φερρυπίν, στην Ουγγαρία έχουμε μια, ε, έχουμε μια σειρά από αυτοφυή δάση, τον οποίο όμως η αποψήλωση ε, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διατεθούν μετά άλλα κονδύλια για να φυτευτούν νέα δέντρα. Και πάλι λίγα χρόνια μετά αρχίζει πάλι η αυθόρμητη αυτή ε, αναδάσωση, η φυσική αυτή αναδάσωση και έχουν εντωμεταξύ χαθεί χρόνια από την εκμετάλλευση αυτή διότι τα, γιατί οι, προ, οι διαδικασίες τις οποίες έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το μεταξύ ε, οδηγούν σε δάση τα οποία αποψηλώνονται. Έχουμε επίσης περιοχές που είναι στο Natura 2000 οι οποίες λόγω της χρηματοδότησης αυτής ή εξαιτίας της χρηματοδότησης αποτρέπουν με τη διαχείριση που γίνεται την αυθόρμητη εμφάνιση δασών. Καλό λοιπόν θα ήταν να γνωρίζουμε τι πράττουμε στην υπόθεση αυτή. Καλύτερη ποιότητα ξύλο και η μεγαλύτερη πυκνότητα δάση ασφαλώ είναι κέρδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το περιβάλλον τη. Οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό. Και επιπλέον υπάρχουν διάφορε περιοχέ απομακρυσμένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή οριακέ ε, φερρυπίν ε, που ε, αποτελούν τις όχθες αυτοκινητοδρόμων όπου θα ήταν σκόπιμο να φυτευτούν δέντρα. Ευχαριστούμε κύριε Γκλατανφέρντερ. Ο κύριος Χόσλιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συμφωνήσω με τόσο υπόθηκαν και από τον εισηγητή και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το να προσδιοριστεί μέσα στο έγγραφο τι σημαίνει δάσος. Δάσος έλεγα εγώ αυθόρμητο ότι είναι ε, αυτό το οποίο εντοπίζει κανεί δέντρα. Όχι, ε, δάσος έχει μια συγκεκριμένη περιγραφή και ορισμό, δηλαδή χρειάζεται πάνω από 10% ε, κάλυψη των εδαφών με δέντρα. Ε, από εκεί και πέρα πρέπει να εξετάσουμε τι είδους, περιβολο... πολιτική θέλουμε για την προστασία των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά δεν αξιολογούνται επαρκώς η ε, θετική, ε, δεν αξιολογείται επαρκώς θετική προσφορά των δέντρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ίσως θα πρέπει να είναι ο πρώτος μας στόχος. Ειδικά στα κράτη της Νότιας Ευρώπης έχει τεράστιο ρόλο διαφύλαξης του κλίματος αλλά και προστασίας των οικοσυστημάτων και Μάλιστα θα επισημάνω μια έκθεση που είχαμε ε, πρόσφατα στην ε, Επιτροπή μας που αναφερόταν στις μεγάλες πυρκαγιές στα δάση στην Νότια Ευρώπη. Με δεδομένο αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα δάση και θα πρέπει να δούμε πολύ πιο προσεκτικά τι σημαίνει όφελος τι καλό μπορεί να προσφέρει το δάσος. Επίσης υπάρχουν διεθνείς προδιαγραφές, συστήματα πιστοποίησης, τα οποία νομίζω μπορούν να αποτελέσουν μια καλή βάση για την ε, εξασφάλιση μιας καλής διαχείρισης των δασών, ενιαίας διαχείρισης. Έχουμε δε ε, ανάγκη να εξετάσουμε και τους πόρους που μπορούμε να αποκομίσουμε από το δάσος και τη διαχείριση της ενέργειας αλλά και την πτυχή της υπερεκμετάλλευσης στον τομέα των δασών. Μπορεί να προσδιορίσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση προδιαγραφές σε ορισμένες περιοχές, ε, όχι λίγες, και υπόθηκε μάλιστα και νωρίτερα, ε, υπάρχουν ε, δέντρα τα οποία δεν ανήκουν στα αυτοφύη ήδη και επηρεάζουν το οικοσύστημα. Θα έπρεπε λοιπόν να ανατρέψουμε αυτήν την τάση και να είμαστε πιο προσεκτικοί στο τι είδο δέντρα φυτεύουμε. Και βέβαια πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, αναπτύξει πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν και την αξιοπιστία τους γιατί όταν υποδεικνύουμε σε τρίτα κράτη τι είδου δέντρα θα πρέπει να φυτεύουν και τι στάση θα πρέπει να τηρούν σε σχέση με τα δάση τους, καλό θα ήταν και εμείς να φροντίσουμε και να προστατεύσουμε τα δικά μας δέντρα και τα δικά μας δάση. Μην κοιτώντα μόνο τον οικονομικό, το οικονομικό όφελος, αλλά και το ουσιαστικό, το περιβαλλοντικό, οικολογικό όφελος. Έτσι λοιπόν αυτό που θα ήθελα να προτείνω εγώ ως τελική ιδέα είναι η προστασία των δασών. Ευχαριστώ Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά από όσα ήθελα να πω ήδη καλύφθηκαν. Σε κάθε περίπτωση το πιο σημαντικό στοιχείο που ήθελα να ακούσω ο συγγετής μας πέραν το ότι συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα μας εξέθεσε είναι το εξή. Θα πρέπει να γίνουν τεράστιες προσπάθειες ώστε οι μέρημνες της γνωμοδότησης αυτής να συνδυαστούν ε, με τις προτεραιότητες ε, που θα προκύψουν από τη γνωμοδότηση για την μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Δεν έχουν κοινοτικοποιηθεί ακόμη τα δάση. Ε, τρέψτε με αυτή την έκφραση. Ξέρουμε ότι τα ευρωπαϊκά δάση είναι πολύ τερογενή μεταξύ τους, πολύ διαφορετικά. Αυτό όμως είναι ένας τομέας που καλύπτεται από το δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ και θα είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα που θα προβληθούν εκεί για τα δάση. Θα πρέπει λοιπόν να εξακολουθήσουμε αλλά και να συνεχίσουμε να ενισχύουμε αυτή τη συνιστόση με έναν υψηλό βαθμό επικουρικότητα για συγκεκριμένε περιπτώσει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω χάρη τη Πορτογαλία, όπω είπε και η συνόδελφο Πατράου Νέβε, έχουμε σοβαρότατα προβλήματα με τι δασικέ πυρκαγιέ. Εδώ έχουμε ζημιέ, έχουμε καταστροφές μάλλον ε, δασικέ, αλλά και ανθρώπινα θύματα. Το 2005, λόγου χάρη, κάτι που το θεωρούσα απίστευτο, έζησα καταιγίδε χωρίς κεραυνούς μάλλον χωρίς να υπάρχει βροχή. Υπήρχαν αστραπές οι οποίες προκαλούσαν απίστευτες πυρκαγιές που λάμβαναν ε, διαστάσεις ε, ασύλληπτες και προκαλούσαν πρικαγιές. Άρα λοιπόν ε, η, τα δάση έχουν ε, περάσει από πολλά στάδια αποψήλωσης ανά τους αιώνες λόγω της ναυπηγίας, της ναυπηγικής μάλλον λόγω της ε, οικοδόμησης των και τι δημιουργίε των δικτύων των σιδηροδρομικών ήταν πολλοί λόγοι που υπήρχε αποψήλωση των δασών, περιορισμό του και οι δασικέ πυρκαγιέ μεταξύ άλλων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν μέρημνα για όλα αυτά τα ζητήματα, για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, για τον περιορισμό τη μείωση τη δασική έκταση. Μέτρα λοιπόν για την προστασία των δασών σε χώρε όπω η δική μου δεν είναι αδιανόητα χωρί μεγάλη δημοσιοδότηση από, εξωτερικά, από εξωτερικές πηγές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η δασική συνιστόσα για όλε τι χώρε και μεταξύ αυτών και για τη δική μου, την Πορτογαλία. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε αυτή την κατεύθυνση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Καπουλασάντος. Κλείνουμε τώρα με τον κύριο Ανιό. Άγνιο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνήθω δική μου αρμοδιότητα είναι να δίνω μια άλλη οπτική γωνία στη συζήτηση. Επειδή λοιπόν ακούσαμε την κλιματική αλλαγή να αναφέρεται στη συζήτηση, τις τελευταίου δύο χειμώνε είχαμε πολύ μεγάλε φαινοπτώσει και τα τελευταία δύο καλοκαίρια είχαμε ελάχιστε, μάλλον πολλέ βροχοπτώσει, 100 μιλιλίτρα μερισίω στη δική μου μόνο περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι και οι γενετικώ οργανισμοί θα επηρεάσουν τα δάση και οι κλιματικέ αλλαγές. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ότι ίσω ένα νέο όρο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα δεν είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά η υπερψύχρανση του πλανήτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλου του συμμετέχοντε. Να δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή, συγκεκριμένα στον κύριο Σούλτ που θα μας ε, εκφράσει τις παρατηρήσεις του και μετά ο κύριος Νικολέσκου. Κύριε Σούλτ. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ηγητές. Αλλά και όλο τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Είδα πολύ ευρύ ενδιαφέρον και ερωτήσεις σε σχέση με την ε, πράσινη βίβλο. Ήθελα λοιπόν να πω ότι το έγγραφο που το έχουμε συντάξει με βάση βέβαια συμβολή και παρατηρήσεις και όλων των εμπλεκομένων, των ενδιαφερομένων ε, παραγόντων έχει και περιβαλλοντική πτυχή αλλά όχι μόνο έχει και άλλες ε, πτυχές του, της χρησιμότητας του δάσους, οποίες ε, δεν αρνούμεθα. Έχουμε επίσης θέματα μέσα στο έγγραφο καταγράψει, γιατί είδαμε από την ανακοίνωση πέρυσι για την προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή ότι υπήρχε τέτοιου είδου ε, ανάγκη και είχαμε πει ότι θα ξεκινούσε μια συζήτηση πρώτα για την ε, συζήτηση και ανταλλαγή απόψε αλλά και ενημέρωση και είπαμε ότι θα πρέπει να ε, ενημερώσουμε τη στρατηγική για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τώρα έχουμε συζητήσει σε συμβουλίου, των ομάδων εργασία δηλαδή, πολιτική προστασία, ακούστηκε το θέμα των δασικών πυρκαγιών, έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση, έχουμε την πράσινη βίβλο, έχουμε μια διάσκεψη ενό του επίπεδου στο, στην Ισπανία την Άνοιξη. Ξεκίνησαμε και δημόσιες διαβουλεύσεις στο τέλη Ιουλίου με 160 τώρα πλέον απαντήσεις στα ερωτήματά μας, τις οποίες απαντήσεις πρέπει να αναλύσουμε. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει. Το Συμβούλιο μας έχει ζητήσει μια δήλωση για τις ε, διαβουλεύσεις αυτές, τον ανοιχτό αυτό διάλογο. Ίσως χρειαστούμε λίγο παραπάνω χρόνο γιατί χρειάζεται με πολύ μεγάλη προσοχή να αναλύσουμε τις πολυάριθμε απαντήσεις που έχουμε λάβει. Και φυσικά δεν χρειάζεται να πω ότι κάθε παρέμβαση υπολογίζεται, σταθμίζεται, αξιολογείται τελό. Επίσης συνεχίζουμε τη μελέτη του, της πράσινης βιβλίου. Χαίρομαι και για τις στάση του Κοινοβουλίου και περιμένουμε και την επόμενη έκθεση που θα συντάξετε διαβεβαιώνοντάς σας ταυτόχρονα ότι είμαστε στη θέσή σας για κάθε τι που ενδεχομένως να χρειαστείτε. Και αν θεωρείτε, πολύ ευχαριστώ να συζητήσουμε απευθείας και με τον εισηγητή διμερός. Όπως είπα, είναι καλός ο σχεδιασμός, θεωρούμε, είναι ευπρόσδεκτο το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για την Πράσινη Βίβλο και προσβλέπουμε στην έκθεση που θα υποβληθεί αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σούλτ και όλους τους ε, συναδέλφους που μίλησαν. Θα δώσω λόγο τώρα στον κύριο Νικουλέσκου για κάποια τελικά σχόλια. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο για τις απόψεις του. Σίγουρα θα λάβω υπόψη τις προτάσεις που κάνατε όταν ολοκληρώσω την σύνταξη της έκθεσης. Ευχαριστώ επίσης την Κομισιόν για τις πληροφορίες που χορηγεί, χορήγησε. Να, υπο, υπογραμμίσω κάτι. Οι περισσότεροι συνάδελφοι προφανώς εκφράζουν ανησυχίες για το μέλλον του δασικού τομέα. Αλλά δεν είναι αυτό το αντικείμενο της έκθεσης. Εγώ θα ήθελα να, να, σας τονίσω ότι η έκθεση αφορά την κατάσταση των δασών. Προφανώς μας ανησυχούν τα τοπικά κλίματα, τα τοπικά δάση, τα δάση σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτό πρέπει να είναι αντικείμενο μιας άλλης έκθεσης ωστόσο. Να σας πω επίσης ότι θα λάβω υπόψη όλες τις απόψεις που ακούγονται εδώ. Αν θέλετε με κάποια τροπολογία να αλλάξετε την έκθεση του ώστε η γνωμοδότησή μας να γίνει πληρέστερη θα τις εξετάσω με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νικουλέσκου. Κλείσαμε τη συζήτηση αυτή και περνάμε στο σημείο 15. Ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την κατάσταση στον ανθοκομικό τομέα να καλωσορίσω τον κύριο πολίτη από την ε, ε, Ιταλική Συνομοσπονδία Γεωργών που θα μας παρουσιάσει την κατάσταση της ανθοκομίας εξ ονόματος του, της Ομοσπονδίας του γιατί συχνά στην Επιτροπή μας, ε, μάλλον σπάνια συζητάμε στην Επιτροπή μας τον τομέα αυτό συνάδελφοι, όμως είναι ένας σημαντικός τομέας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτη παραγωγός καλοπιστικών φυτών παγκοσμίω. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη κοινοτικών επιδοτήσεων για να επιβιώσουν οι ανθοκομικές εταιρείες της Ευρώπης. Όμως ε, με την κρίση στον τομέα των τροφίμων γενικότερα έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και στον τομέα των ανθοκομικών. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να δούμε και σε το επίπεδο της Επιτροπής μας το όλο αυτό ζήτημα. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο στου υπευθύνου των πολιτικών ομάδων, θα ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής και έπειτα οι ενδιαφερόμενοι θα θέσουν τα ερωτήματά του. κύριος Πολίτη, ευχαριστώ κύριε Μεκάστρο και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές που βρίσκονται σήμερα εδώ για να με ακούσουν. Εκπροσωπώ τους ε, ανθοκαλλιεργητές της Ιταλίας που εκπροσωπεί μαζί μου και η κυρία Μαριάντζελα Κατάνιο η ίδια ανθοκαλλιεργήτρια υπεύθυνη εκ μέρους της δικής της περιφερειακής οργάνωσης. Οργανώσαμε πρόσφατα στο Σαρέμο μία ημερίδα προβληματισμού, ημέρα και ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα του τομέα αυτού, για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Ο ανθοκομικός τομέας στην Ευρώπη καταγράφει κέρδο 20 δις ευρώ. Είναι λοιπόν οικονομικού βάρους που δεν μπορεί να παραμεληθεί. Ιδίως ό,τι αφορά την χώρα μου, την Ιταλία, η εταιρείε ενθοκομικέ είναι 36.000 με 100.000 εργαζομένους. Ο ενθοκομικό τομέα, ανέκαθεν ήταν μέρο τη ε, ελεύθερη αγορά, τη ανοιχτή αγορά και δεν είχε οικονομική στήριξη ούτε συγκεκριμένη διοργάνωση, μια κοινή οργάνωση αγορά, όπω συμβαίνει σε άλλου τομεί, με άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα. Υπάρχει μάλιστα μια διαδομένη προκατάληψη που κατατάσσει τον τομέα αυτό στους πλούσιους και θεωρεί ότι καταγράφονται κέρδη χωρί καμία πολιτική στήριξη. Στο παρελθόν σίγουρα είχαμε λιγότερα προβλήματα σε σχέση με άλλου τομεί. Όμω, τώρα ο τομέας πλήττεται από την παγκόσμια κρίση με συρρήκνωση τη ζήτηση, αλλά και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που και των αρνητικών συνεπειών που είχαν προκύψει ήδη πριν την εκδήλωση της παγκόσμιας κρίσης. Αυτό αφορά όλου τους ανθοκόμους στην ε, Ευρώπη, όχι μόνο τους ε, Ιταλούς. Ιδίω ε, στην καλλιέργεια των καλοπιστικών φυτών, με περιορισμό τη έκταση καλλιέργεια, 26% μόνο στην Ιταλία, αλλά γενικότερα όλων των παραγωγικών περιοχών στην Ευρώπη. Εδώ αυτό συμβαίνει ενώ οι εισαγωγέ από τι τρίτε χώρε συνεχώ αυξάνονται. Αυτή τη στιγμή το 74% των ε, καλοπιστικών φυτών που ε, είναι αντικείμενο πορεία στην Ευρώπη προέρχονται από τρίτες χώρες. Σήμερα οι Ευρωπαίοι παραγωγοί πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα επίπεδο ανταγωνισμού ανυπόφορο αν σκεφτούμε ότι η μέση τιμή του τριαντάφυλλου πέρσι μειώθηκε κατά 50% από 50 λεπτά σε 35 λεπτά. Μεγάλες απώλειες λοιπόν για τον τομέα μας και αυτό με κάποιες ε, ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες ευνοϊκές για τις τέτοιες χώρες, την Νότια Αμερική και την Αφρική. Και ταυτόχρονα την απουσία περιβαλλοντικών ε, προδιαγραφών για την τοπική παραγωγή καθώς και πολλά κίνητρα για να φύγουν ε, κάποιες εταιρείε και να πάνε να παράγουν σε τρίτες χώρες. Να εγκαταστήσουν εκεί δηλαδή την παραγωγή τους. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί λοιπόν έχουν προβλήματα και ω προ το εργατικό δυναμικό, αλλά αντιμετωπίζουν και τι δυσκολίε προμήθεια ενέργεια και τι περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ που είναι πολύ αυστηρέ. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε κατά πόσον εδώ οι αναπτυξιακέ ε, επιδοτήσει. Ε, και οι δασμολογικές ελαφρύνσεις των τρίτων χωρών είναι εύστοχες. 50% των καλοπιστικών φυτών έρχονται στην αγορά μας με μηδέν δασμούς. Έτσι λοιπόν έχουμε δυσκολίες με τον ανταγωνισμό που πολλές φορές γίνεται αθέμητος και άδικος για τους ευρωπαίους παραγωγούς. Ακόμη υπάρχουν και επιδοτήσεις για τη μετακίνηση εταιριών, κάτι που δεν επιτρέπει την τοπική ανάπτυξη και άνθηση του τομέα αυτού. Ε, οι Ευρωπαίοι επίση χάνουν πολλού από του φυσικού του πόρου με την υποβάθμιση του, όπω ε, αυτών των υδάτινων πόρων. Και αυτό πλήττει τι τοπικέ κοινότητε. Τα προβλήματα αυτά, βάσει των ιδιαιτεροτήτων που κατέγραψα, αλλά και βάσει τη κόπα, θα πρέπει να έχουμε εδώ ε, συγκεκριμένα με εργαλεία απλά που να στηρίξουν το τομέα μα. Να θυμίσω ορισμένα. Αναθεώρηση κοινοτικών πολιτικών πρόσφατα ε, προέβλεψε ότι θα δίνονται στήριξη μόνο σε εταιρείε. Θα υπάρχουν λοιπόν επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο σε εταιρείε που θα επιτρέπουν την ευρωπαϊκή ανάπτυξή τους. Αλλά αυτό δεν έχει καμία λογική εφόσον ουσιαστικά ε, εταιρείε αυτές <clears throat> καταλήγουν να μετακινούνται και στηρίζουμε τους τρίτους παραγωγούς. Επίσης, οι, ευρωπαϊκέ οι ευρωπαϊκές εταιρείες τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να ωφεληθούν από τις διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με τη χρήση των παρασιτοκτόνων σε τρίτες χώρες και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Χρειάζονται έλεγχοι αποτελεσματικοί και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Γιατί υπάρχουν πολλές ε, βλαβερές ουσίες και σε, αυτές, σε αυτά τα προϊόντα. Στους καταναλωτές λοιπόν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα αποφύγουν την εισαγωγή και διάδοση νόσων και παρασίτων. Θα πρέπει να προβλέψει υγειονομικέ υπεχρώσεις η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και για τα εισαγόμενα προϊόντα, όπω ακριβώ για τα ευρωπαϊκά όταν εξάγονται στι εξωκοινωτικέ χώρε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αμοιβαιότητα στην ε, εμπορευματοποίηση των ε, τροφίμων ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει επίσης ο τομέας της ανθοκομικής να συμπεριληφθεί ο σκέλος στο σύνολο της κοινή αγροτικής πολιτικής μετά το 2013. Θα πρέπει ο τομέας αυτός να μην θεωρείται απομονωμένος από τους υπόλοιπους της γεωργίας. Επίσης, η παγκοσμιοποίηση της κοινωτικής νομοθεσίας θα πρέπει να, προ βλέψει και διευκολύνσεις για τη χρήση της ε, για τη χρήση του πετρελαίου. Ε, επίσης θα πρέπει η παραγωγή ανθοκομική και καλοπιστικών φυτών να υποφεληθεί από τις προσπάθειες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να λάβει υπόψη περιβαλλοντικέ μερίμνε, αλλά και για την ενεργειακή εξοικονόμηση. Θα πρέπει λοιπόν να κλείσω λέγοντα ότι όλα τα μου τη Ομοσπονδία, αλλά και οι Ευρωπαίοι Ανθοκόμοι συνολικά, θα πρέπει να ε, βρεθούν σε τέτοιε συνθήκε ώστε να, απλώ να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν, να φτιάχνουν λουλούδια δεν είναι αναγκαστικά ένα είδος πολυτελείας ε, τα λουλούδια, αλλά ένα σύμβολο της ομορφιάς της φύσης. Και είναι ένα, ένα σύμβολο ευημερία και καλής ε, διαβίωσης για όλους μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πολίτη. Όντω θα είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση, διότι ο ανθοκομικός τομέα αντιμετωπίζει προβλήματα και αυτό αφορά πολλέ εταιρείε στην Ευρώπη. Όπω είπατε έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Τα προβλήματα λοιπόν στα οποία δώσατε έμφαση είναι πρακτικά συγκεκριμένα και υπάρχει πραγματικά πτώση στον, στις επενδύσεις στον τομέα αυτό. Να συζητήσουμε τώρα πριν ακούσουμε τον κύριο Γέρογκαν από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Ο κύριο Ταραμπέλα, έχετε στο λόγο. Μάρκ. Ευχαριστώ. Άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο πολίτη και τα λόγια του πραγματικά ενισχύουν τους φόβους μας όταν μιλούμε, μίλησε για την τιμή του τριαντάφυλλου που μειώθηκε διότι υπάρχουν σε άλλες υπήρους πιο ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες προφανώς Νότιος Αφρική, Αφρική γενικά, Νότιος Αμερική επίσης μίλησε και για την Κολομβία τα περισσότερα τριαντάφυλλα που μας πουλάνε στα εστιατόρια προφανώς από εκεί έρχονται. Τόνισε επίσης ε, και άλλα ζητήματα. Περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί κανόνες ε, που διέπουν την παραγωγή. Πριν από κάποια χρόνια είχα μιλήσει με Κολομβιανούς ε, συνδικαλιστές του κλάδου της ανθοκομείας οι οποίοι είχαν έρθει για να καταγγείλουν, τότε δεν ήμουν ευρωβουλευτής ακόμα, τις συνθήκες παραγωγής που ήταν σκανδαλώδεις. Λέμε προστασία του περιβάλλοντο. Μην ξεχνάτε ότι είναι άνθρωποι που δουλεύουν γυμνοί, χωρίς μάσκες, με παρασυντοκτόνα. Το προσδόκιμο ζωή του ζωής τους είναι 35 βία. Η ζωή τους χάνεται. Ε, τότε είχαμε συνάψει μια συμφωνία όταν θέλουμε να συνάψουμε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με χώρε όπω αυτή, η Κολομβία δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε και τέτοιε διαστάσει. Δεύτερον, από, υπάρχουν κανόνες, αποτελεσματικοί κανόνες κα, ε, παραγωγής. Ε, η, η Γερμανία είχε ξεκινήσει νομίζω ένα σήμα παραγωγής που τηρεί τα περιβαλλοντικά κοινωνικά ε, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές. Δεν ξέρω τι έγινε μετά βέβαια. Μπορούμε να προβλέψουμε διότι έχουμε και μαζικές εισαγωγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο λουλουδιών από εκεί. Υπάρχουν έλεγχοι των ε, κανόνων παραγωγής από αυτή τη διάσταση. Γιατί σε μια χρονική στιγμή με κάτι, με κάτι τέτοιες δυνατότητες, σωστά το έθεσε ο κύριος Πολίτη, μιλάμε, μπορεί να μιλήσουμε για αφέμιτο ανταγωνισμό. Μπορεί να μην μπορούμε να εμποδίσουμε το ευδείχνε εμπόριο, αλλά ασκήθηκαν τουλάχιστον πιέσει προ τι χώρε αυτέ για να βελτιώσουν τι ε, ε, τους, τις συνθήκες ε, παραγωγής τους. Γιατί μετά ερχόμαστε και φωνάζουμε στις ε, ευρωπαϊκέ εταιρείε που σηκώνουν και φεύγουν και πηγαίνουν ε, τις επιχειρήσεις του αλλού. Ευχαριστώ. Σίγουρα θα απαντήσει η Επιτροπή. Έχουμε και εκπρόσωπο της Επιτροπής του κ. Τζενάτα, ο οποίος ε, μπορεί να απαντήσει. Η κυρία Γέγκλε έχει ζητήσει το λόγο. Η Ελίζαμπετ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλύφθηκα από τον Σαλφα Ταραμπέλα σε μεγάλο μέρος των όσων είχα να πω. Δεν μπορώ παρά να υποστήριξω τα ερωτήματα που διατυπώνει. Καλό βέβαια να συμφωνούμε στις, ε, στους προβληματισμούς και τους λογισμούς μας από όλες τις ομάδες. Δεν θέλω να επισημάνω. Το τομέα είναι πολύ σημαντικός. Και εγώ ως Γερμανίδα επιβεβαιώνω και το γεγονό ότι σε μια προσφατή μας λίστα επίσκεψη ανθοκομικό και εκδήλωση επεσήμανα αντελήφθη μάλλον τα ίδια προβλήματα και για το εργατικό δυναμικό και για το κόστος ε, των προστατευτικών προϊόντων και επίσης εδώ με μια πρόσθετη ερώτηση όπως είπε ο Μαχ σε ποιο βαθμό προχωρεί η εναρμόνιση ή έχει προχωρήσει η εναρμόνιση στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ποιο βαθμό θα ήταν χρήσιμο να εναρμονίσουμε τον τομέα αυτόν. Και πρέπει να πω ότι με πολύ υπερηφάνεια άκουσα ότι μέσα στις συνθήκες ελεύθερης αγοράς έχει μπορέσει να επιβιώσει και με, καλές, με καλή ανταγωνιστική σχέση ο χώρος ανθοκομείας, αλλά τώρα ίσως χρειάζεται πλέον κάποια υποστήριξη, ενίσχυση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως και την προσδοκά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει περισσότερο τι είδους προβλέψεις έχει κάνει, πώς έχει συζητήσει την κατάσταση αυτή, τι θα μπορούσαμε να έχουμε υπόψη για το μέλλον του τομέα αυτού στην Ευρώπη ολόκληρη, τι θα βοηθούσε ή τι θα μπορούσε ενδεχομένω να αποβεί εις φάρος ε, του τομέα. Ο, κύριος έχει συζητήσει το λόγο. Η κυρία Ντελάνγκε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πολίτη και εγώ για τις θέσεις του. Νομίζω ότι η κρίση όντως υπάρχει παντού. 7% των εκμεταλλεύσεων στην χώρα μου ε, σταμάτησαν τη δουλειά τους, ενώ η ανθοκομεία είναι πολύ ισχυρό κλάδος ε, στην Ολλανδία. Δεν συμφωνώ ωστόσο με κάποιες από τις προτάσεις που ακούστηκαν. Η λύση είναι, πρέπει να ζητήσει, οι λύσεις που προτείνουν οι Ιταλικές ε, οργανώσεις είναι μια προσέγγιση αλλά υπάρχουν και άλλες προτάσεις λύσεων από άλλους οργανισμούς. Η μετακίνηση επιχειρήσεων δεν γίνεται μόνο προς τα έξω, γίνεται και προς τα μέσα. Είναι ενιαία αγορά, αλλά υπάρχουν ε, οι εθνικές αρχές έχουν χρηματοδοτήσει την μετακίνηση επιχειρήσεων ε, στο εσωτερικό της Ένωσης. Βλέπουμε ότι ο κλάδος θέλει υποστήριξη. Μπορεί αυτή η υποστήριξη να, από τα διαφορετικά ταμεία ωστόσο να αποβεί αντιπαραγωγική, Παρεπιπτόντως το λέω αυτό. Σε ό,τι αφορά τη λύση που πρέπει να βρούμε θα πρέπει να στηριχθεί στα ισχυρά σημεία του κλάδου. Φερρυπίν, προώθηση, ενέργεια. Στον κλάδο αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας. Υπάρχουν θερμοκήπια που έχουν ε, ουδέ, που είναι ουδέτερα που έχουν στην παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα ή που εξοικονομούν ενέργεια. Πρόκειται για έργα που πρέπει να χρηματοδοτηθούν και να ενισχυθούν. Καινοτομία. Άλλο σημαντικό στοιχείο. Ως Κοινοβούλιο εμείς προσπαθούμε να προασπίσουμε τις ε, ε, εξαιρεσει για τους δικαιούχους ε, ευρεσιτεχνιών. Όσοι ωστόσο έχουν τέτοιες ευρεσιτεχνίες πρέπει να μπορούν να προχωρήσουν. Έχουν λοιπόν, υπάρχει, ωστόσο υπάρχουν οι εξαιρέσεις για τους δικαιούχους που, τους, που εμποδίζουν τους επιχειρηματίες να εκμεταλλευτούν τα νέα ε, ευρήματα. Θα ζητούσα από τους συναδέλφους να επανεξετάσουν την προσέγγιση αυτή. Θα πρέπει να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την κοινοτομία. Συμφωνώ ότι υπάρχουν ότι πρέπει να υπάρχουν ε, αντίστοιχες απαιτήσει για την τοπική παραγωγή και τις εισαγωγές. Καλό είναι να υπάρχουν και ευρωπαϊκά λογότυπα, αλλά αυτό ε, δεν είναι το βασικό. Το λουλούδι είναι ένα προϊόν μάζας. Κατά την άποψή μου, αυτό που σίγουρα δεν πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε μια νέα πολιτική με μέτρα που θα αντιμετωπιστούν ή θα θεωρηθούν ως προστατευτικού χαρακτήρα. Αναφέρθηκε ότι πρέπει να ε, καταργηθούν οι προτιμήσεις, οι προτιμησιακές συμφωνίες. Ωστόσο, τέτοιες συμφωνίες είναι αυτές που ε, βοηθούν τις φτωχότερες χώρες και τους φτωχότερους στις φτωχότερες χώρες. Θέλουμε να σταματήσουμε να βοηθάμε στις Δεν νομίζω ότι η ανθοκομεία πρέπει να είναι το μέσο ή το εργαλείο κατάργησης των προτιμήσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μία συζήτηση ζωηρή, ουσιαστική, για την αναζήτηση λύσεων. Οι λύσεις αυτές πρέπει να ξεκινήσουν από το ότι ζούμε στον 21ο αιώνα και από το ότι ε, έχουμε μια σειρά ισχυρών στοιχείων. Ε, Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες ε, των ανθοκαλλιεργητών. Ε, σωστά τα είπε και ο κύριος Ταραμπέλα που μίλησε για την ανάγκη υιοθέτηση ε, κανόνων παρόμοιων και στις χώρες εκτός της Ένωσης. Δεν θέλουμε να έχουμε νέους περιορισμούς ωστόσο. Καλύτερα θα ήταν να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο το, τους κανόνες, ε, τους περιβαλλοντικούς και, εργατικούς, και εργασιακούς κανόνες κάτω από τους οποίους ε, παράγονται τα λουλούδια στις άλλες ε, περιοχές του κόσμου. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε σαφώς το εξής. Ό,τι εισάγεται στην Ευρώπη, στα λουλούδια και σε όλες τις άλλες πολιτικές, πρέπει να γίνεται με βάση ε, τις, ε, τα ίδια επίπεδα, τις ίδιες απαιτήσει που ισχύουν για την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο πρέπει να πούμε και αυτό θα βοηθήσει όλους όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανθοκομείας. Βεβαίως, είναι σε κάποιες χώρες ε, πολύ σημαντικός κλάδος. Νομίζω τα λουλούδια αποτελούν από τα σημαντικότερα προϊόντα εξαγωγής της Κένια. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε ούτως ώστε να εφαρμόζονται οι ίδιες συνθήκες παντού. Δεν είναι προστατευτισμός αυτός. Οι περιβαλλοντικές ε, προϋποθέσεις ισχύουν όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για τις τρίτες χώρες. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπει ο κλάδο στην ε, κοινή γεωργική πολιτική. Μπορεί να το χρειάζεται να το συζητήσουμε σε κάποια χρονική στιγμή. Ε, συμφωνώ μαζί σα. Είναι ένα σημαντικό κλάδος με μεγάλη σημασία για τις μικρές επιχειρήσεις που πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Ο κλάδος της ε, ανθοκομίας είναι κλάδος που παλιά έδινε πολλές θέσεις εργασίας. Άλλαξε κάτι διάρκεια της, των τελευταίων ετών, εξαρτάται ιδίω από κατανάλωση ενέργειας. Αυτά τα δύο στοιχεία εξηγούν νομίζω την μετακίνηση της ανθοκομείας από την Ευρώπη σε χώρες ε, εκτός Ένωσης που έχουν εργατικό κόστος μικρότερο και καλύτερο, καλύτερες κλιματικές συνθήκες που οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Βεβαίως αυτό γίνεται και σε άλλες υπήρους. Ε, ζητάμε, ε, συζητάμε στο Κοινοβούριο τις εξελίξεις, τι πρέπει να κάνουμε για την αλλαγή του κλίματος αν εξετάσουμε την, το ενδεχόμενο εισαγωγή ενό φόρου διοξιδίου του άνθρακα στο εσωτερικό, ο κλάδο τη ανθοκομεία σίγουρα θα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και θα, ήταν, θα είχε θετικά αποτελέσματα γι' αυτόν. Η ανθοκομία στην Ευρώπη πληρώνει το τίμημα της επαγγελματική ανεπάρκειας και σε, ιδίως σε εμπορικό επίπεδο έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις που ανταγωνιζόντουσαν επί μακρόν η μία την άλλη που παρήχαν παρόμοιο προϊόν και προσπαθούσαν να αντισταθούν στις μασικές εισαγωγές. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον κλάδο πρέπει να τον παρατρύνουμε να κάνει καλύτερη εμπορική οργάνωση της παραγωγής και της πρόθεσης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκλάτφελντερ. Ευχαριστώ. Όταν είχαμε τη, την κρίση του Ισλανδικού ηφαιστείου και δηλαδή είχα μείνει εδώ και δεν μπορούσα να πάω σπίτι μου, άκουγα στο BBC, είδα στο BBC μάλλον, ένα ντοκιμαντέρ για τις πολύ δύσκολες ε, συνθήκες που, κάτω από τις οποίες δούλευαν ε, που αντιμετώπιζαν τότε οι ανθοκόμοι, η παραγωγή λουλουδιών στην Αφρική που δεν μπορούσαν να φέρουν τα λουλούδια του στην Ευρώπη. Θα ερχόντουσαν αυτά στην Ευρώπη, τα προϊόντα δηλαδή, μέσα σε μικρά σε ψυγιάκια θα ερχόντουσαν στην Ευρώπη. Σε φορτηγά δηλαδή που σε, ε, μεταφορικά μέσα που ψύχονταν. Το ίδιο συμβαίνει και με, πολλές, ε, και με πολλά λουλούδια στην Ευρώπη. Κατά την άποψή μου δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τους λίγους ε, πόρους ε, ορυκτών καυσίμων που διαθέτουμε σε τέτοια μέσα. Δηλαδή ε, κλιματιζόμενα οχήματα που μεταφέρουν λουλούδια. Θα έπρεπε να δούμε ποιο είναι το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα των λουλουδιών που μεταφέρονται. Ευχαριστούμε κύριε και ο κύριος Μποβέ. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω τον εκπρόσωπο των Ιταλών παραγωγών, τον κύριο Πολίτη. Ε, τον καλωσορίζω και τον χαιρετίζω συναδελφικά. Για το θέμα αυτό της παραγωγής ανθέων υπάρχουν πολλά προβλήματα σχετικά. Πρώτα απ' όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Είναι πολλά τα χημικά που χρησιμοποιούνται σήμερα. Έχουμε ζητήματα ρήπανση και σε αυτό το τομέα. Και αυτό πρώτα απ' όλα πλήττει του εργαζομένου τη νοσοκομεία. Δεύτερο πρόβλημα. Η περιοχή του Νότου και τη Δυτική Γαλλίας αυτή τη στιγμή έχει θυσιαστεί τελείω στο όφελο της ε, παραγωγή Στην περιοχή των Άλπαιων, κοντά στην ε, θάλασσα, παραθαλάσσια δηλαδή, και νοτίως ε, ο τομέας αυτό καταστρέφεται. Μιλάμε για εκατομμύρια εκτάρια αυτή τη στιγμή που είναι εγκαταλελειμμένα. Εάν λοιπόν θέλουμε οι ανθοκόμοι να έχουν ένα εισόδημα και να μην αντιμετωπίζουν την, τον αθέμητο ανταγωνισμό, ε, πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τι θα κάνουμε. Μιλήσαμε προηγουμένω για την Κένια. Εγώ επισκέφτηκα πριν από λίγα χρόνια θερμοκήπια και μια εγκατάσταση παραγωγή αντέων στην Κολομβία. Η κατάσταση ήταν δραματική και ήταν ε, συγκρίσιμη και μάλλον με τη χρήση των ε, λιπασμάτων ε, υπήρχε τέ, πολύ ψηλό ποσοστό ασθενειών. Υπάρχει λοιπόν ο φόρο για την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, αλλά όπω λέμε και για την παραγωγή των προϊόντων από ζώα, πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο σεβασμό από. Εφόσον υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο ελάχιστο αριθμό προδιαγραφών, θα πρέπει να σκεφτούμε και εμεί τι κάνουμε με τα εισαγόμενα προϊόντα. Δεν μπορεί να εισάγουμε προϊόντα από χώρε που δεν σέβονται καθόλου την υγεία των εργαζομένων του και φέρνουν προϊόντα που μπορεί να έχουν βλάψει την υγεία του. Ευχαριστούμε τον κύριο Μποβέ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή. Ο κύριος Βέρουγκαν. Και έπειτα ίσως και ο κύριος Ντενάντας από τη Γενική ΣΑΝΚΟ. Eh, eh, ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα να περιγράψω τα όσα κάνουμε στην πολιτική της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας για αυτόν τον τομέα. Στη Γενική Διεύθυνση λοιπόν ασχολούμαστε με την παρακολούθηση της αγοράς των καλοπιστικών αθέων και θεωρούμε ότι είναι σημαντικέ επαφέ μα με του εκπροσώπου του τομέα, μαζί με τι συμβουλευτικέ επιτροπέ που συστηματικά συνέρχονται. Παρακολουθούμε λοιπόν συστηματικά την κατάσταση στον τομέα αυτό και βλέπουμε τι προβλήματα υπάρχουν. Ο τομέα αυτό συμπεριελήφθη το 2007 στην κοινή οργάνωση αγορά, την ενιαία οργάνωση αγορά, αλλά δεν προβλέπονται ειδικά μέτρα για αυτόν. Ωστόσο, στον ε, τομέα αυτό υπάρχουν κονδύλια που προβλέπονται από διαφημιστικά προγράμματα και υπάρχει κοινοτική συμβολή κατά 5%. Ο σκοπός είναι να δείξουμε τα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών προϊόντων ιδίως ό,τι αφορά την ποιότητα της μεθόδους παραγωγής, τις υγειονομικές συνιστώσεις και την ε, βάλλοντος πέραν των κονδυλίων λοιπόν αυτών για τα διαφημιστικά προγράμματα. Στηρίζουμε βάσει του δευτέρου πυλώνα της κοινή αγροτικής πολιτικής στον τομέα στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης, των προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου. Σε ό,τι αφορά την πορεία του τομέα, την οποία σφιγμομετρούμε συστηματικά, βλέπουμε ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δυσχερή α, ήδη από το 2009. Για μια μακρά περίοδο σημειώνονταν αύξηση, συστηματική αύξηση της παραγωγής στην Ευρώπη από το 2000 έως το 2009 με μια αύξηση περίπου 20%. Όμως η αύξηση αυτή επιβραδύνθηκε το 2009 με μείωση 1,2%. Ταυτόχρονα με την αύξηση της παραγωγής για μια μακρά περίοδο Είδαμε ότι και οι επιφάνειες αυξήθηκαν κατά 7% σε, αυτήν, σε αυτά τα 9 χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση στις κατοχώρες. Όπως υπόθηκε πρόσφατα, αυξήθηκαν και οι εισαγωγές τα τελευταία δύο χρόνια, με εξαίρεση την περσινή χρονιά. Μειώθηκε, σημειώθηκε μείωση 6,5%. Όπως αυξήθηκαν όμως οι εισαγωγές, ταυτόχρονα αυξήθηκαν και οι εξαγωγές. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στον τομέα αυτό. Ειδού λοιπόν πως έχουν τα πράγματα όπως τα έχουμε καταγράψει εμείς. Όπω είπα προηγουμένω, δεν προβλέπονται ειδικά μέτρα πέραν των διαφημιστικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων ανάπτυξη τη υπαίθρου. Αυτή είναι η κατάσταση και το νομικό πλαίσιο όπως δημορφώνεται σήμερα. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ την κυρία Γερόγκαν. Βέργαν. Ε, προφανώς τα αριθμητικά δεδομένα είναι αυτά που μα αναφέρατε. Περιμένουμε απαντήσει στι ερωτήσει μα βεβαίω δεδομένου ότι η σε αυτή κατάσταση είναι πραγματικότητα. Είναι πολύπλοκοι και κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει το ζήτημα τη αμοιβαιότητα που τόσε φορέ το έχουμε θίξει στην Επιτροπή μα για άλλα γεωργικά προϊόντα, για άλλε μορφέ παραγωγή και υπάρχουν και όλε αυτέ οι δυσκολίε ω προ τον ανταγωνισμό που κάποιε φορέ γίνεται αθέμητος Κάποιε ε, φορέ έχουμε ίδιοι διώξει την παραγωγή μας από την Ευρώπη και μετά φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους ίδιους του παραγωγούς μας στην Ευρώπη. Να προσθέσω κι εγώ κάτι. Εκτός αν θέλει να παρέμβει και το άλλο μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι, ναι. Ο κυρίος Γενάτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να στην ερώτηση που έθεσε ο κύριος Μποβέ και το ζήτημα της, το θέμα του του ανταγωνισμού. Και προηγουμένως στο ερώτημα του προηγούμενου βουλευτού για τους ελέγχους στο μεταποιημένο προϊόν. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω ότι στο πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων με τους εταίρους μας, με τα άλλα κράτη. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε και τις συνθήκες συνεργασίας, αλλά και να αντιληφθούμε καλύτερα τι συμβαίνει ακριβώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα τρίτα κράτη ως προς τη χρήση των συζανιοκτώνων. Σε αυτές τις μέρες λοιπόν επαφές πάντοτε επισημαίνουμε και το τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είδους νομοθεσία έχουμε ως προς τη χρήση των ζυζανιοκτώνων, όποια και είναι αυτά, και τους ελέγχους που έχουμε εμείς για να περιορίζουμε τις δυσμανείς επιπτώσεις, επιβλαβείς επιπτώσεις αυτών των ζανιοκτώνων. Επίσης υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα και επιμένουμε μια άλλη πτυχή, ε, τη σχετική με την πνευματική ιδιοκτησία των προϊόντων, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο εξασφαλίζεται η προστασία για τα φυτά και ιδιαίτερα και συμπεριλαμβανομένων μάλλον και των διακοσμητικών ε, φυτών ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ε, ορίζει άλλωστε και η Διεθνή Σύμβαση υπό του 1991, προστασία δηλαδή των διαφορών ειδών φυτών. Τα κράτη αυτά με τα οποία συνομιλούμε πολύ συχνά δείχνουν ενδιαφέρον. Θέλουν να ενταχθούν και τα ίδια στην διεθνή αυτή σύμβαση και προσπαθούμε να τα πείσουμε φυσικά πάντα. Και έτσι έρχομαι πρόεδρε στο ζήτημα του αθέμη του ανταγωνισμού, όπου πιστεύω θα πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη προσπάθεια να ενημερώνουμε και τους δικού μας παραγωγούς και δικαιούχου. που είναι συχνά μικρέ και μεσαίες επιχειρήσεις. Πριν να εξάγουν λοιπόν, καλό θα είναι να είναι ενήμεροι για την προστασία του προϊόντος που εξάγουν του προστατευόμενου προϊόντος που εξάγουν, έτσι ώστε οι είναι σε θέση και να βοηθούν ε, στην αναπαραγωγή και τον και στα κράτη αυτά και σε περίπτωση επανεξαγωγής των προϊόντων αυτών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον να έχουν τη δυνατότητα να, ασκήσουν τα δικαιώματά τους επί των προϊόντων αυτών που θα μπορούσαν διαφορετικά είτε να πολλαπλησιαστούν κατά τρόπο απατηλό, είτε να οδηγήσουν σε παραποιήσεις στα κράτη εκείνη τα οποία δεν αναγνωρίσουν ακόμη την προστασία της ε, φυτικής παραγωγής. Σε αυτό θα ήθελα να ε, επισημάνω την προσοχή σας. Να επιστήσω την προσοχή σας σήμερα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει να παρέμβει. Το πρόβλημα παραμένει. Θα δούμε τι πρωτοβουλίες θα αναλυφθούν και μαζί με τους συντονιστές θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε προς την σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ λοιπόν τον πρόεδρο του πολίτη και την ΚΟΠΑ και την ε, ΣΥΑ και εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας. Δεν υπάρχουν άλλα σημεία στην εμμυρίσια διάταξη. Απλώς να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι τη Δευτέρα στις 11 Οκτωβρίου στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ όλους σας. Λίγη συνεδρίαση.